Uh, so good afternoon everybody. I'm sorry we're running slightly late this afternoon. Καθυστερήσαμε λίγο. Καλώς ήρθατε. Έχουμε τεχνικά θέματα της ενιαίας αγοράς. Αρχίσαμε ήδη με τη μελέτη αντικτύπου για τις εγκρίσεις αγροτικών και βιομηχανικών οχημάτων. Τώρα όμως, ο κύριος Παντσέρη θα κάνει σχετικές τροπολογίες και μετά έχουμε και τροπολογίες για τις μοτοσυκλέτες. Και υπάρχουν και ορισμένα τα οποία άπτονται και των δύο. Ω συνήθω έχουμε και ισχυρή εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης του επιχειρήν, κυρίως με τον κύριο Μαρτίνο Παρόντα, που παρακολουθεί το θέμα αυτό από την αρχή. Ας αρχίσουμε λοιπόν την συζήτηση. Χωρίς περισσότερες λοιπόν εισαγωγές θα παρακαλέσω τον κύριο Παντσέρη να κάνει την παρουσίαση του θέματος καθώς και των τροπολογιών του και μετά θα περάσουμε σε ένα γύρο των σκιωδών εισηγητών. Ο κ. Μάντερς είναι παρόν, εγώ είμαι σκιωδός εισηγητής ομάδας μου, η κυρία Ριούλε. Σόντι και η Σαφίνη ακόμη δεν είναι παρόντες. Είσαι ο κ. Σφάπ, που δεν παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, θα φροντίσει ο σκιώδης συγητής του να είναι παρόν όταν θα έρθει η ώρα. Κύριε Παντσέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, ο στόχος της πρότασης είναι να ορίσουμε μία σειρά από κανόνες, εναρμονισμένους κανόνες, για δασικά και γεωργικά οχήματα, για να μπορέσουμε να εγγυθούμε τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να ξεχνάμε την οδική ασφάλεια, την προστασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Η πρόταση, όπως επίσης και την επαγγελματική ασφάλεια, είναι πολύ σημαντική η πρότασή μας, για να μπορέσει να συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα του, του, του κλάδου, Η παρούσα έκθεση είναι το αποτέλεσμα πόλων διαβουλεύσεων που είχαμε με τον ε, κλάδο, χρήστες, ε, συνδικάτα, μηχανικούς κλπ. Και ήταν μια διαδικασία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα που μου επέτρεψε να διατυπώσω μια έκθεση που ελπίζω ότι θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη αλλά και στη φιλοδοξία του να έχουμε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για το θέμα. Κατά τις εργασίες διαπιστώσαμε ορισμένα σημεία τα οποία θα ήθελα να σας υποβάλω σύντομα ελπίζω. Πρώτα οι προδιαγραφές τεχνικής ασφάλειας σε σχέση με την οδηγία για τις μηχανές. Δεύτερον, η συμβατότητα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και με, τους, ε, με τις συμφωνίες σχετικά με την ομολογοποίηση. Επίσης, ε, για τα θέματα συντήρησης ε, των οχημάτων, επίσης για τα κίνητα για τα side by side και τα επί τροχών ε, οχήματα και τρίτον για τις προδιαγραφές ασφάλειας και οι σχέσεις με την οδηγία για τα μηχανήματα. Θέλει η Κομισιόν να βγάλουμε τα τρακτέρ και τα δασικά μηχανήματα από την οδηγία για τις μηχανές και αυτό για να μειώσει τις νομικές πράξεις που αφορούν στα τρακτέρ και να προβλέψει την απλούστευση ο αποκλισμός των ε, βασικών και γεωργικών ε, ελκυστήρων από την οδηγία καλύπτονται από τους όρους της οδηγίας για τις μηχανές και για να μπορέσουμε να αποφύγουμε το νομικό κενό. Σήμερα η Κομισιόν αξιολογεί όλα τα ρίσκα τα οποία ρυθμίζονται σήμερα από την οδηγία για τις μηχανές και προβλέπει να τα μεταφέρει στον τωρινό κανονισμό. Πρόκειται για μία δούλια που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στην προνομοθετική φάση και στα άρθρα 7 και 8 της πρότασης θα έπρεπε να προβλέπονται οι συγκεκριμένες προδιαγραφές της οδηγίας για τις μηχανές. Η κατεξουσιοδότηση πράξης δεν μπορούν να ορίζουν καμία νέα προδιαγραφή, καμία νέα διάταξη, αλλά πρέπει να θεσπίζουν την εφαρμογή των αποφασισμένων διατάξεων. Για την λειτουργική ασφάλεια και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εγώ καθορίζω τρόπολογική τροπολογίες οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται από την πρόταση, δεν εξετάζονται από την πρόταση της Κομισιόν. Θα ήθελα να εξεταστούν αυτές οι διατάξεις ούτω ώστε να μπορέσουμε στα άρθρα 7 και 8 και στο παράρτημα 1 του κανονισμού να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι οδηγίες ούτω ώστε να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες ελκυστήρων. Έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες ε, που θέλουν να προσαρμόσουν τις διατάξεις αυτού του κανονισμού στη διάταξη 778 του 2008 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό πλαίσιο για την εμπορευματοποίηση των προϊόντων, ούτως ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή και η εκτέλεση αυτού του κανονισμού. Αυτές οι διατάξεις διευκρινίζουν τον ρόλο των οικονομικών χρηστών όσον αφορά στην εποπτεία. Το post-market, δηλαδή μετά τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά και τον έλεγχο των προϊόντων που εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Ενισχύονται επίσης οι διατάξεις σχετικά με οργανισμούς που θα μπορούσαν να αναλάβουν κατανάθεση από τα κράτη-μέλη ελεγκτικές αρμοδιότητες και να περιφρουρήσουν την εφαρμογή της οδηγίας. Λαμβάνονται υπόψη και οι προσπάθειες της παράλληλης ομάδας ε, εργασίας του Συμβουλίου για την Τεχνική Εναρμόνιση και για την ε, ομολογοποίηση των διαφόρων οχημάτων μεταξύ των οποίων των τρικύκλων και των τετρακύκλων. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι αυτά τα οποία οδηγούν στο να έχουμε πολλές τροπολογίες για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων. Σήμερα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη ως προς τη συντήρηση και αυτό λόγω των ηλεκτρονικών ε, στοιχείων των μηχανών που δεν μπορούν να επισκευαστούν με την παραδοσιακή μηχανική. Χρειάζονται για την επισκευή πλήρης πληροφορίες για την παρεμβολή στα ηλεκτρονικά συστήματα. Οι χρήστες έχουν ε, οι χρήστες ε, σήμερα ε, ρυθμίζουν την επισκευή των μηχανημάτων τους στις βάση των συμφωνιών που έχουν οι πολιτές με τις αντιπροσωπείες και τα συνεργεία. Υπάρχει λοιπόν μια μονοβολιακή κατάσταση. Θα έπρεπε να προσέξουμε ούτως ώστε η διαδικασία να μην παρακολύει την πρόσβαση στην αγορά των ανεξαρτήτων συνεργείων. Πρόκειται για ανεξάρτητα μηχανικά συνεργεία τα οποία βρίσκονται σε ε, απομακρυσμένες περιοχές ε, της Ένωσης και που μπορούν να συμβάλλουν στην ε, επισκευή και μικροεπισκευή των μηχανών αυτών. Επίσης πρέπει να προσέξουμε και τις ε, αντιφατικές, τις συζητήσεις που έχουμε σχετικά με την υψηλή τιμή των, των ανταλλακτικών. Θα πρέπει να δούμε, να περιφρουρήσουμε τους ανεξάρτητους ε, χρήστες οι οποίοι δεν έχουν τα μέσα στη διάθεσή τους για να προασπίσουν τα συμφέροντά τους. Η πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες θα πρέπει να είναι πλήρης ε, για όλους ε, στο όνομα της προστασίας ε, του ανταγωνισμού και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για τα κινούμενα οχήματα θέλω να πω ότι η Κομισιόν στην πρόταση της έχει μια νέα κατηγορία που είναι, η μη είναι τα τροχοφόρα τα οποία όμως δεν κυκλοφορούν σε δρόμους. και θα πρέπει η Κομισιόν να εξετάσει ποια είναι τα εθνικά ζητούμενα για αυτού του τύπου τις μηχανές και να προσαρμοστεί. Εμείς πιστεύουμε ότι στην θέλουμε μάλλον στην εισήγησή μας, στην έκθεσή μας να αποκλείσουμε τα μηχανήματα που εντάσσονται στην κατηγορία Α1 και καλούμε την Κομισιό να υποβάλει μία ειδική πρόταση για αυτού του τύπου τα μηχανήματα. Για τα οχήματα side by side και τα 4x4 είναι, είναι οχήματα που τα χρησιμοποιούμε και στο δασικό τομέα και στη γεωργία. Γι' αυτό θεωρήσαμε να συμπεριληφθούν στον ε, κανονισμό μας. Αυτά τα οχήματα που χρησιμοποιούνται όμως κυρίως για οδική κυκλοφορία και για ψυχαγωγία έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ελκυστήρες, από τα τρακτέρ και θα έπρεπε να ε, ενταχθούν στην ομολογοποίηση της, ε, των οχημάτων της κατηγορίας μη. Θα πρέπει να έχουμε διαφορετική και απαιτήσει ε, για τα υπηρεσιακά 4x4 τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Εγώ θα ήθελα να γίνει παράλληλη συζήτηση για την ένταξη των οχημάτων αυτών στην κατηγορία λάμδα παράλληλα με τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, αναμένοντας ε, και τη σχετική μελέτη της Κομισιόν για τα οχήματα side by side, για να δούμε σε ποια κατηγορία θα πρέπει να εντάξουμε αυτά τα οχήματα. Έχουμε σημαντικές, ε, πολλές μάλλον τροπολογίες τεχνικού χαρακτήρα που θέλουν να διευκρινίσουν τεχνικές πτυχές και θέλουν να διασφαλίσουν και τη μεγαλύτερη σύνοχη του κειμένου. Αυτό εξηγεί και το μεγάλο αριθμό των ε, τροπολογιών. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι η έκθεση αναλύει τα θεμελιώδη ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εξεταχθούν προσεκτικά στην έκθεση. Πρόκειται για σημαντική δουλειά για να μπορέσουμε να συζητήσουμε στην Επιτροπή επικοδομητικά Περιμένω τις προτάσεις των συναδέλφων. 27 Σεπτεμβρίου λίγη η προθεσμία στις 12 για την κατάθεση των τροπολογιών. Και συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Θέλαμε να έχετε επαρκή χρόνο για να μπορέσετε να καλύψετε ενδελεχώς όλα τα σημεία. Βεβαίως ε, δαπανίσατε πολύ χρόνο για να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα για θέματα ζωτικής σημασίας. Θα ήθελα οι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο για θέματα που κάλυψε που δεν κάλυψε ο κύριος Παντζέρη. Σφάμπ. Εγώ θα μιλήσω, λέει ο πρόεδρος, εκ μέρους της ομάδας μου. Και οι άλλοι μπορούν επίσης. Και μετά ο κύριος Μαρτίνο. Ευχαριστώ. Πρώτα θα δηλώσω ότι κολλείεται η κυρία Σαρτόρη. Βλέπω όμως γνωστά πρόσωπα στην γραμματεία και αυτό με ικανοποιεί γιατί θα ήθελα εγώ να είμαι επανεξέτασε Η επανεξέταση αυτή τη οδηγία που είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επιτυχη. Μιλώ τώρα εξ ονόματο τη κυρία Σαρτόρη και ευχαριστώ τον κύριο Παντσέρη για τι λύσει για πολλά λεπτομερή θέματα που έχουν αρκετή, αρκετά περίπλοκο χαρακτήρα. Χαίρετε κύριε Σαρτόρη, ιδίω για τι προόδου που έχει επιτελέσει τώρα η έκθεση σε όλου του προβληματικού ω τώρα τομεί. Ο μεγάλο αριθμό τροπολογιών που έχουν υποβληθεί, όπω ανεμένετο, θα οδηγήσει σε τροποποίησει βέβαια σε διάφορε παραγράφου. Πρώτο σύντομο σχόλιο τη κύρια Σαρτόρη αναφέρεται σε πέντε θέματα, σε πέντε θέματα συγκεκριμένα. Πρώτα, θετική συνεργασία μεταξύ εισηγητού και σκιωδών εισηγητών, που θα οδηγήσει στον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των δύο τμήματων, ε, των δύο νομοθετών δηλαδή. Δεύτερο, κύριε Σαρτόρη, συμφωνεί με τον εισηγητή ότι η κατηγορία ΟΥ, δηλαδή κινητά μηχανήματα, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, διότι είναι απαραίτητο εδώ να γίνουν οι εξαιρέσεις αυτές, επειδή δεν προκύπτουν οι ίδιοι κίνδυνοι από την χρήση των μηχανών αυτών. Επίσης τώρα η εξαίρεση των μικρών οχημάτων παντουδακού εδάφους που λέγονται γουρούνες ε, στην κοινή ελληνική. Το προτείνει αυτό επίσης η κυρία Σαρτόρη για την κατηγορία λάμδα, L, θα προτείνει και άλλες τροπολογίες η κυρία Σαρτόρη. Μετά η κυρία Σαρτόρη, αγαπητέ κύριε Παντσέρη, επανέρχεται στο θέμα του κεφαλαίου 16 Εάν δηλαδή οι ελκυστήρες, τα τρακτέρ, θα τύχουν τις ίδιες μεταχείρισεις όπως τα κλασικά ε, οχήματα, αυτοκίνητα. Εδώ υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις από πλευράς της ομάδας μας, αν είναι δηλαδή σκόπιμο να υπαχθούν στην ίδια μεταχείριση. Η κυρία Σαρτόρη θα συνδιαλεχθεί και πάλι με την ομάδα, πάντως θα υποβάλει σχετικές τροπολογίες. Δηλαδή, οι ελκυστήρες να μην έχουν την ίδια μεταχείριση όπως τα υπόλοιπα αυτοκίνητα οχήματα. Εμείς βεβαίως θέλουμε οι αγορές να μην ανοιχτέ και ιδίω για τα συνεργεία επισκευών. Αυτό είπαν άλλωστε και οι ενδιαφερόμενοι στην διαβούλευση, ότι υπάρχουν δυσκολίες σχετικά με την συντήρηση των διαφόρων δικτύων συνεργείων επισκευών, διότι δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό, πολύ απλά. Γι' αυτό λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα θα υποβάλουμε ε, τροπολογία η οποία θα ζητεί διαφορετική μεταχείριση των δύο αυτών κατηγοριών οχημάτων. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την περαιτέρω συνεργασία και συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάντερς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντσέρη. Η εκθεσή του είναι αρκετά περίπλοκη. Και εγώ προτιμώ που είναι κανονισμός και όχι οδηγία. Αυτή είναι και η σωστή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Συμφωνώ με το ότι οι ελκυστήρες δεν έχουν τις ίδιες απαιτήσει όπως τα αυτοκίνητα. Τα είπε αυτά ο κύριος Σβάμπ. Όμως εάν κυκλοφορούν στους δημόσιους ε, στους δρόμους θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση διότι, διότι τότε βέβαια προκαλούν και παρόμοιους κινδύνους. Βέβαια λένε οι ενδιαφερόμενοι ότι τα τρακτέρ τα χρησιμοποιούμε στα χωράφια. Ναι, αλλά για να φτάσουν στα χωράφια πρέπει να περάσουν από το δικό δίκτυο. Τώρα, για την 44. Νομίζω ότι εδώ ζητείται η καταχώρηση Δεν γνωρίζω αν αυτό είναι ορατό εκ των έξω. Σε ορισμένες χώρες είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αριθμός κυκλοφορίας στο πίσω μέρος του οχήματος, αλλά σε άλλες χώρες δεν είναι απαραίτητο, δεν προβλέπεται υποχρεωτικά. Νομίζω ότι χρειάζεται, νομίζω ότι χρειάζεται πανευρωπαϊκή ρύθμιση, γιατί τότε θα είναι ε, σαφές να μπορεί αμέσως να αντιληφθεί κανείς δηλαδή αν πρόκειται για καταχωρισμένο όχημα ή όχι. Εγώ θέλω να υπάρχει λοιπόν αριθμός κυκλοφορίας, καταχώρηση κυκλοφορίας δηλαδή, στο πίσω μέρος του οχήματο. Και τέλος, το πιο σημαντικό, Βεβαίω μπορεί κανείς να πει ότι ε, δεν υπάγεται εδώ, διότι είναι τεχνική έκθεση. Αλλά θα πρέπει να απαιτήσουμε ορισμένες ε, προϋποθέσεις ασφαλείας και από πλευρά οδηγών ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο για την εκπαίδευση των οδηγών. Αυτά τα οχήματα, ελκυστήρες κλπ. γίνονται όλο και μεγαλύτερα και όλο και ισχυρότερα. Και βλέπω καμιά φορά νεαρά παιδιά 16 ετών να τα οδηγούν. Όταν μιλούμε λοιπόν για απαιτήσει ασφαλεία, ο οδηγό είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξουμε. Αυτά ήθελα να πω για την ώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάστηκε και επανεπεξεργάστη την πρόταση και έχει κανείς την εντύπωση ότι τα σκέφτηκε πραγματικά όλα. Θερμός έπαινος λοιπόν, οι πτυχές που με ενδιαφέραν εμένα, η ολόκληρη αυτή η κατηγορία U, Υπάρχουν προβλήματα με άλλες ρυθμίσεις που ισχύουν στον τομέα αυτό. Εγώ βρίσκω την πρότασή του ευφυή και σκόπιμη. Καθώς επίσης και αυτά τα quad πάλι μου έστειλαν επιστολές και μου λένε ότι δεν θέλουν να υπαχθούν στην κατηγορία L, λάμδα, αλλά θέλουν να παραμείνουν στα, στην κατηγορία των τρακτέρ. Βεβαίως συχνά τα οχήματα αυτά δεν χρησιμοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Οι περίφημες γουρούνες λοιπόν. Εγώ θεωρώ τότε ότι οι απαιτήσει ασφαλείας και εκπομπών καυσερίων κτλ. θα πρέπει να ε, συμμορφώνονται και για αυτά τα οχήματα δηλαδή με αυτές των υπολείπων αυτοκινήτων. Για το πλαίσιο τώρα των ε, συντηρήσεων, να εξετάσω λίγο και το θέμα των εκπομπών. Ομολογώ ότι δεν είχα την ευκαιρία να μπω στις λεπτομέρειες, θα το πράξω, αλλά έχω εκ πρώτης όψεως την εντύπωση ότι πραγματικά σκέφτηκε ο κ. Παντσέρη όλες τις λεπτομέρειες και το εκφράζω τις ευχαριστίες μου και το σεβασμό μου. Θα μιλήσω κι εγώ ως σκιώδης συγητής. Θα επανέλθω στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Πραγματικά είναι εξαιρετικά τεχνική η έκθεση και είναι σπάνιο η συγητής να έχει εγκύψει τόσο σοβαρά σε τέτοιο τεχνικό θέμα και να έχει συντάξει 292 τροπολογίες. Λίγα σχόλια μόνο για να απαντήσω στα όσα είπατε. Το θέμα της επικαλύψεως με την οδηγία περί μηχανημάτων. Είναι γνωστό το πρόβλημα αυτό, τα είπε και ο κύριος Σφάπ. Έχουμε κάποια τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση του θέματος. Όσο περισσότερη πίεση ασκηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κάποιες ξεκάθαρες λύσεις, τόσο καλύτερο. Η νέα κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα βεβαίως όσον αφορά τη διαδικασία επιτροπολογίας μας αναγκάζει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να φροντίσουμε ο κανονισμός αυτός να έχει επαρκές πεδίο εφαρμογής. Νομίζω ότι χρειάζεται να το προωθήσουμε γιατί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα λόγω της ασάφειας αυτής της επικάλυψης με την οδηγία περί μηχανημάτων. Πρέπει αυτές οι δύο να ε, ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο κείμενο που, με τρόπο που να μην αφήνει κενά. Η μόνη ανησυχία τώρα είναι ότι είναι ευρύτατο το φάσμα των τεχνολογιών από τις πλέον απλές μέχρι τις πλέον περίπλοκες. Και το ερώτημα για μένα είναι εάν σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο και η τελευταία λεπτομέρεια ή και η τελευταία τεχνική λεπτομέρεια ενός ε, ελκυστήρα που έχει και ηλεκτρονικά ε, συστήματα ε, διευθύνσεως και που μπορεί να κοστίζει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Είναι απαραίτητο να είναι ρυθμισμένο με τον ίδιο τρόπο όπως και ένα απλό μηχάνημα. Νομίζω ότι από αυτού θα χρειαστεί να αναζητήσουμε τις συμβουλές πραγματογνωμόνων. Στα γεωργικά μηχανήματα ασφαλώς και ενσωματώνονται τώρα πολύ περίπλοκες ηλεκτρονικές τεχνολογίες και θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό το δρόμο για το μέλλον. Φροντίζοντα όμως να είναι επαρκώς καλυμμένοι. Βασικό λοιπόν με τις βασικές, συμφωνώ μάλλον με τις βασικές αρχέ σα, αλλά θα ήθελα αυτά τα πράγματα να είναι όλα καλυμμένα. Σε ό,τι αφορά τι ρυθμιστικέ απαιτήσει για εξαιρούμενα μηχανήματα κινητά μηχανήματα. Τι απαιτήσει δηλαδή για την χρήση τους επί του οδικού δικτύου. Δεν είναι, είναι απαράδεκτο να έχουμε τέτοιες παραλλαγές από χώρα σε χώρα. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σφαιρικότερα. Αυτό που προτείνεται νομίζω είναι πράγματι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Και υποστηρίζω τη γραμμή που προτείνεται. όσον αφορά τον αποκλεισμό των κινητών μηχανημάτων. Αλλά θα παρακαλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγύψει το δυνατόν συντομότερο και να έρθει σε επαφή με του κατασκευαστέ μηχανημάτων. Όσον αφορά τα οχήματα παντοδαπού εδάφου, καλά κάνουμε και το, χρησιμοποιούμε, και το ε, συζητούμε ταυτόχρονα με την έκθεση του κ. Βάντε Κάμπ και χαίρομαι που τον βλέπω παρόντα εδώ, διότι είναι κάτι το οποίο εμένα τουλάχιστον με έχει ανησυχήσει μέχρι τώρα έκανα ορισμένες προτάσεις και τροπολογίες για την έκθεση Van de Kamp που έχουν ως στόχο να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή υποκατηγορία για αυτά τα λεγόμενα quad γουρούνες όπου εγώ σημειώνω ότι υπάρχουν ορισμένα ξεχωριστά χαρακτηριστικά μηχανημάτων τέτοιων που χρησιμοποιούνται για αγροτική χρήση και που ε, τα καθιστούν πολύ διαφορετικά από άλλα τα οποία χρησιμοποιούνται για χρήση επί του δρόμου. Είναι διαφορετικές απαιτήσει και θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι κατασκευαστές οι οποίοι παράγουν οχήματα για χρήση εκτός δρόμου να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση. Για παράδειγμα με την εγκατάσταση διαφορικών στα μηχανήματα αυτά και ούτω καθεξής μία από τις προτάσεις Βαντεκάμπ νομίζω ότι καλύπτει τις απαιτήσεις αυτές. Μπορούμε τώρα να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί και μαζί μας αλλά και με τους κατασκευαστές για να εξασφαλιστούν να εξασφαλιστεί τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας και περιβαλλοντικών. Χωρίς ωστόσο να οδηγηθούμε σε μειονέκτημα των ε, κατασκευαστών μηχανημάτων εκτός ε, δρόμου. Αυτά είναι τα βασικά που ήθελα να πω ως σκιώδης. Και ευχαρίστω τώρα να ανοίξω την συζήτηση, αν θέλει κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Κανείς. Ah, yes, I just wanted, Mrs. Violet reminded me, I just wanted η κυρία Βάιλερ μου υπενθύμισε ότι θα πρέπει να καλωσορίσω τους μαθητές του σχολείου Richard Μίλλερ από την Φούλντα. Είμαι βέβαιος ότι θα έχετε τρομερό ενδιαφέρον για γεωργικούς ελκυστήρες, αλλά θα μιλήσουμε και για μοτοσυκλέτες και για κουάντ. Και είμαι βέβαιος ότι αυτά θα σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Κύριε Μαρτίνο, θέλετε να δώσετε μια πρώτη απάντηση στις προτάσεις του κυρίου Παντσέρη. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα και σας ευχαριστώ διότι δίνετε τη δυνατότητα στην Επιτροπή να σχολιάσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παντσέρη για τις εργασίες του, για την εργασία του, Μιλάμε για τεχνικά ζητήματα, δεν είναι εύκολο το ζήτημα και θεωρούμε ότι το σχέδιο έκθεσης του ε, ασχολείται με όλα τα επιμέρους στοιχεία. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι δεχόμαστε την προσέγγιση του. Καλωσορίζουμε λοιπόν το γεγονός ότι η έκθεση λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις μεταβλητές της αγοράς, καθώς και τις άλλες προτάσεις που υπάρχουν επί τάπητος. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την εποπτεία της αγοράς και να ε, προωθήσουμε το συντονισμό. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον εισηγητή γιατί ακριβώς ε, με αυτό το ζήτημα ασχολήθηκε. Ως προς την ε, προσέγγιση για, τις ε, κινητές, για τα κινητά μηχανήματα, θεωρώ ότι τα στοιχεία είναι πολύ σωστά. Για τα, για τα οχήματα αυτά. Στην μελέτη αντικτύπου είδαμε ποιες είναι οι επιλογές των κατασκευαστών. Δηλαδή, κατά πόσο η οδηγία ανταποκρίνεται στην οδική ασφάλεια. Αυτό θα το κάνουμε όμως για τα οχήματα και μηχανήματα που αφορούν γεωργικές εργασίες ή δασοκομικές. Κάπως προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά Πιστεύω ότι η προτινόμενη προσέγγιση ζητώντας από την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτό το θέμα συνεκτικά θεωρούμε ότι αντιμετωπίζεται πολύ σωστά. Σε σχέση με τα ATV θεωρούμε ότι προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη όλες τις επιμέρους πτυχές έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μηχανήματα και οχήματα τα οποία σχεδιάζονται ειδικά και πολλούνται. Δεν είναι προϊόντα αναψυχής. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, ιδιαίτερα και να δώσουμε μεγάλη προσοχή. Κύριε Σέρμαν, μιλήσατε και για τη δική σας πρόταση. Θεωρούμε ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανταποκριθούμε. Θα πρέπει λοιπόν να καλύψουμε όλων των ειδών τα οχήματα και να λάβουμε υπόψη συγκεκριμένες προαπαιτήσεις για τις υποκατηγορίες που αφορούν γεωργική καθαρά χρήση. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για μία επιλογή στην οποία θα προσδώσουμε μεγάλη σημασία. Μιλάμε για τα οχήματα side by side καθώς και άλλα. Έχουμε αναλάβει μία μελέτη για να λάβουμε υπόψη και επιπρόσθετα στοιχεία. Σε σχέση με επισκευές και τα συναφή, γνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα των ελκυστήρων, καθώς και των δασοκομικών οχημάτων και μηχανών. Θεωρούμε σημαντικό να έχουμε όλες τις πληροφορίες μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας και θα πρέπει να συντονιστούμε όπως κάναμε και σε άλλους τομείς, δηλαδή να δούμε ποιες είναι συγκεκριμένες ανάγκες των ελκυστήρων. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτές τις υποδείξεις έτσι ώστε να φτάσουμε στη σωστή ισορροπία σε σχέση με τους γεωρικούς ελκυστήρες. Ένα πιο λεπτό ζήτημα που αφορά την οδηγία περί και ίσως εδώ υπάρχει επικάλυψη. Θα ήθελα να πω ότι εδώ λάβαμε υπόψη τα δεδομένα που μας αναφέρεται καθώς και του κυρίου Σβάπ. Το 2006 είχαμε αποφασίσει να αποφύγουμε την επικάλυψη μεταξύ των δύο νομοθετικών κειμένων. Όμως η πρόταση που έχουμε δεν είναι το τέλος της διαδικασίας. Βρισκόμαστε στο μέσο της διαδικασίας γιατί με τις προτάσεις που ήδη εγκρίθηκαν πέρσι είχαμε περιλάβει και ορισμένους κινδύνους οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μιλούσαμε για τους έξι κινδύνους που θα πρέπει να μας αποσχολήσουμε στα πλαίσια των προδιαγραφών και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης. Πρόσφατα αναθεωρήσαμε τους κανονισμούς για τα γεωργικά μηχανήματα και ελκυστήρες. Άρα θεωρούμε ότι δεν υπάρχει την οδηγία περί μηχανημάτων και μηχανών. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ενημέρωση αυτών των δεδομένων ανατύπω Θα ήθελα επίσης να σας ανακοινώσω ότι έχουμε οργανώσει για τις 14 Σεπτεμβρίου μία άτυπη ομάδα εργασίας για τους γεωργικού, γεωργικούς ελκυστήρες, έτσι ώστε να αναλύσουμε και να δούμε ποιες είναι οι απαιτήσεις ασφάλειας και για, ιδιαίτερα ως προς την αναεπάγγελμα ασφάλεια, επαγγελματική ασφάλεια. Θεωρούμε λοιπόν ότι στην ομοθεσία αυτή πλαίσιο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να τα εντάξουμε όλα σωστά με τις ε, κατεκτέλεση πράξεις. Και όπως είπατε δεν ε, κάνουμε μία διαδικασία copy-paste με βάση το κείμενο, το προϋπάρχον κείμενο, απλώς ε, προσπαθούμε να δώσουμε μία έγκριση ανατύπω έτσι ώστε να είμαστε ακριβείς ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις που θα πρέπει να ενταχθούν στην νομοθεσία. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να καλύψουμε αυτόν τον τομέα με βάση την ασφάλεια οχημάτων για να έχουμε ορισμένα συγκεκριμένα στοιχεία για να μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε και να επικαιροποιήσουμε τις απαιτήσει αυτές, τις προπαιτήσει αυτές. Θα ήθελα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε σχέση με τις προαπαιτήσει στην οδηγία μηχανημάτων, διότι δεν συνάδει απόλυτα με την ε, νομοθεσία που αφορά την έγκριση τύπων. Σας ευχαριστώ. Μας δώσατε σαφείς απαντήσεις και θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία έγκρισης. Κύριε Παντζέρη, θα θέλατε να απαντήσετε σε, αυτά που είπε ο κύριος Μαρτίνο και να μας πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και άλλα τυχόν σημεία που έχουν ανακύψει. Από τη συζήτηση έχετε το λόγο. Grazie. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ όλους σας, τους και όντις εισηγητές και την Επιτροπή για όλα όσα είπατε και για την κρίση σας στη δουλειά μου. Συμφωνώ με πολλούς από σας, διότι εμείς ακολουθήσαμε ένα δρόμο ο οποίος για να εγγυθεί υψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας, ασφάλεια στον χώρο της εργασίας, ασφάλεια των μηχανημάτων και προστασία του περιβάλλοντος, χρειάζεται μία διαδικασία έγκρισης τύπου σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να λαμβάνεται η υπόψη το κόστος ωφέλεια, κυρίως για τις ΜΜΕ, αλλά αυτό με, ιδιαίτερα, με, με ιδιαίτερες προπτικές Σύμφωνο, Πρόεδρε, ότι πρέπει να βρούμε την σωστή ισορροπία για να αποφύγουμε την επικάλυψη μεταξύ οδηγιών. Θέλουμε να ασκήσουμε πίεση για να μπορέσουμε στο μέλλον να έχουμε ένα πιο συνεκτικό και ισορροπημένο πλαίσιο. Οι απαντήσεις της Κομισιόν τίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Όσον αφορά το θέμα των 4x4, εγώ στην έκθεσή μου αναφέρω προτάσεις. Και αυτό που αναφέρατε εσείς, η πρόταση που κάνατε, νομίζω ότι επίσης ευσταθεί για να μπορέσουμε να βρούμε την καλύτερη λύση. Φυσικά, είμαι στην διάθεση των σχεδόν εισηγητών μέχρι την προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 27 Σεπτεμβρίου στις 12. Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου εγώ είμαι έτοιμος να συζητήσω με όποιον το θέλει. Ευχαριστώ. So, just on the time Ως προς το χρονοδιάγραμμα θα ήθελα να το δούμε ένα λεπτό προθεσμία υποβολής τροπολογιών 27 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Στη συνέχεια, 17 Οκτωβρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες, θα ψηφίσουμε στις 22 Νοεμβρίου στην Επιτροπή και αυτό σημαίνει ότι στην Ολομέλεια μάλλον θα ψηφίσουμε το Φεβρουάριο του 2012. Αυτό ηχεί σαν να βρίσκεται πολύ μακριά, αλλά είναι μεγάλος όγκος εργασίας. Συμφωνεί ο εισηγητής, εντάξει και η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ για, ε, για την εργασία σας. Πάμε στο δεύτερο θέμα, βασικό θέμα, που έχει προχωρήσει αρκετά αφορά τα δίκυκλα και τρίκυκλα, καθώς και τετράκυκλα. Ο κύριος Βαντεκάμπ ήταν πολύ απασχολημένος με το δίκυκλο του το καλοκαίρι. Έχουμε γύρω, γύρω στις 200 τροπολογίες. Στις 6 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε. Γι' αυτό θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να δούμε τις τροπολογίες και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε συμβιβασμούς και μετά θα το ε, δούμε με τους σκιώδες. Ο κύριος Μάντερς είναι εδώ, Ρούλε, ο υποφαινόμενος, η κυρία Στάιλε. Ναι, θα ασχοληθείτε και εσείς με το θέμα. Η κυρία Στάιλε θα ασχοληθεί με θέματα δικύκλων σήμερα. Βάντεκαμπ, πείτε μας λοιπόν, τι πορεία ακολουθήσατε τον Αύγουστο με το ε, δίκη και ο κύριος Μαρτίνο θα μας απαντήσει. Πάντε καν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι όλοι σας θα περάσατε εξαιρετικές διακοπές. Βέβαια, εγώ είχα ένα πρόβλημα, αν δεν είχα τη μοτοσυκλέτα μου, δεν θα είχα πέσει την προηγούμενη τρίτη. Βέβαια, έχω αρχίσει και συνηθίζω στις πτώσεις τώρα τελευταία. Και βέβαια, στο κεφάλι, το κεφάλι μου δεν έπαθε τίποτα, αλλά τα πόδια μου ναι. Στο, στην ιστοσελίδα, στα αγγλικά, λέτε, γράφετε ότι εγώ είμαι ένας, ε, ότι και μοτοσυκλετιστής. Όμως εγώ είμαι ευρωβουλευτής. Βέβαια, ως ευρωβουλευτής ακολουθώ το σωστό, το, το σωστό δρόμο, πρόεδρε ως μοτοσυκλητιστής λίγο λιγότερο. Εγώ πέρασα το καλοκαίρι μου για να σοβαρολογήσουμε τώρα κύριε Πρόεδρε, μελετώντας τις τροπολογίες. Και κατέληξα ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Έχουμε τρεις τάσεις σε αυτή την Επιτροπή. Την βασική τάση Βάντερ που φυσικά έχει και τη σαφή πλειοψηφία. Μετά έχουμε την έκθεση Ριουρβερσφάλ. που είναι η γραμμή, της, ε, η γραμμή από αριστερά και του Χάρμπορ που από δεξιά εκφράζει και αυτός ε, την γραμμή Εκφράζει λοιπόν έλεγα ο Χάρμπορ την δεξιά γραμμή που έχει και αυτή την πλειοψηφία της. Είχαμε συναντήσεις με τους ε, σκιώδεις εισηγητές και θα στείλω ένα σημείωμα στον συντονιστή μου λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε έτσι. Για τα εκτός ε, δρόμου οχήματα Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έλεγε ο συνάδελφος Παντζέρη. Η Ιαπωνέζικη βιομηχανία μου στείλε προτάσεις για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Θα κοιτάξω να τα λάβω υπόψη μου. Αλλά αυτό σημαίνει ότι και στην έκθεση Παντζέρη θα πρέπει να συμπεριληφθούν ορισμένα από αυτά τα στοιχεία. Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε καλά ε, σε, καλά αποτελέσματα για τον συμβιβασμό. Δεύτερη τροπολογία για την on-board διαγνώσεις. Ο κύριος Βέστφαλ ε, ε, λέει ότι και ο τελευταίος μοτοσυκλητιστής θα πρέπει να είναι τροφοδοτημένος. Πρόεδρε, έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα για τις ε, εκπομπές. Οι κύριοι Ρούλε και Βεστφάλεν θέλουν πολύ πιο αυστηρές απαιτήσεις. Εσείς όμως, εμπνευσμένος από την Βρετανική κυβέρνηση που έκανε μία ανάλυση κόστους ωφέλειας για την περίπτωση, εσείς ε, διατηρήσατε μία συνέπεια στις τροπολογίες σας. Εντελώς αντιφατική με την άλλη πρόταση και δεν ξέρω πώς μπορούμε να βρούμε συμβιβασμό. Άλλο πρόβλημα που έχω και φαντάζομαι δεν θα βρούμε συμβιβασμούς είναι το ηλεκτρικό αποδήλατο. Η κυρία Ρούλε παρουσίαση σε τροπολογίες αλλά δεν υπάρχει εδώ καμία πλειοψηφία ενόψη. Και δεν το λέω δηλαδή αρνητικά αλλά πιστεύω ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε λύση. Η Κομισιόν ε, ε, το έχει στην καρδιά της ε, το θέμα των τεχνικών προδιαγραφών για το ηλεκτρικό ποδήλατο. Πρέπει και αυτό λοιπόν το θέμα παραμένει <coughs> ανοιχτό. Και το χρονοδιάγραμμα Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας για το θέμα των εκπομπών. Τα τεστ. Τα τεστ στις μηχανές που έχουν ξεπεράσει τις 50.000 χιλιόμετρα, πώς μπορούν να, να αντέξουν στο χρόνο. Εσείς ε, Εσείς ε, ε, εξετάσατε φαντάζομαι το τεστ ε, Καλιφόρνια, αλλά αυτό δεν ισχύει. Τα μεγάλα προβλήματα λοιπόν είναι τα ATV, τα OBV, οι εκπομπές, <coughs> τα ηλεκτρικά ποδήλατα και η διάρκεια των μηχανών. Θα μπορέσετε να απαντήσετε τώρα. <coughs> Αλλά νομίζω δεν αναφερθήκατε ειδικά στο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων, ABS δηλαδή, που υπήρχε κάποια διαφωνία. Εσείς τι ακριβώς θέλετε να σας απαντήσω. Νομίζετε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Ναι, υπήρχαν κάποιες διαφορές απόψεων. Νομίζω δεν αναφερθήκατε απλώς στο ABS. Αυτό είναι δική μου παράληψη, πράγματι, κύριε Πρόεδρε. Διάφορα ε, ζητήματα που στρέφονται γύρω από το ABS και το CBS, που είναι τρόποι δηλαδή τροχοπέδησης των οχημάτων, Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι επιθυμούν όλα τα δίκυκλα οχήματα να έχουν το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος, άλλοι που θεωρούν πως όχι. Ε, και πρέπει βέβαια να γίνει κάποια προσπάθεια συνδιαλλαγής μεταξύ των δύο απόψεων. Ας κάνουμε ένα πρώτο γύρο συζητήσεως. Θα ακούσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μπορέσετε να επανέλθετε. Και βεβαίως θα συναντηθούν οι ε, σκιώδεις την επόμενη εβδομάδα. Η κυρία Στάιλερ. Κολλείται σήμερα η κυρία Βέστφαλ που είναι η κυρίως αρμοδία και σας ζητήσει συγγνώμη και με παρακάλεσε να μεταφέρω τα σχόλιά, τα σχόλιά της, αν συμφωνείτε. Η κυρία Βέσφαλ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και με τις τροπολογίες της, διότι θεωρεί ότι τα, συστήματα αντιμπλοκαρίσματος θα πρέπει να είναι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τα EBS με μόνη εξαίρεση δίκυκλα κάτω των 50 κυβικών εκατοστών και που δεν έχουν ταχύτητες κάτι τέτοιο. Δηλαδή μοτοποδήλατα στην πραγματικότητα. Μπορούν λοιπόν να μειωθούν τα ατυχήματα με τη χρήση των συστημάτων αυτών. Ελπίζει ότι θα μειωθεί και το κόστος Αυτό είναι, εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα της κυρίας Βέστφαλ και ελπίζω ότι ο κύριος Βαντεκάμ θα μπορέσει να το λάβει υπόψη του. Δεν έχετε τίποτε άλλο, άλλο σχόλιο. Καλώς. Κύριε Μάντερς, εσείς. Έτσι παίρνει και στην έκθεση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαντερκάμπ για τη δουλειά του. Το ABS και οι εκπομπές είναι πράγματα πολύ τεχνικά και θα πρέπει να τα αφήσουμε στους εμπειρογνώμονες. Αυτό που μας καίει είναι να είναι ασφαλείς οι μοτοσυκλέτες. Και το κοινοβούλιο πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να είναι ασφαλείς οι μοτοσυκλέτες, γιατί μέχρι σήμερα δεν το είναι. Και ο συνάδελφος Ροσφόρ αυτό θέλει. Ε, και αυτό ισχύει φυσικά και για τα τρακτέρ και τα βασικά οχήματα. Στην, στο όλο σύστημα ασφάλειας, στο κεντρικό σημείο θα πρέπει να είναι ο οδηγός. Και ο κύριος Βαντερκάμπ ίσως θα έπρεπε να κυκλοφορεί με τρίκυκλο, διότι αν πέφτει ο κύριος Βαντερκάμπ με όλη την εμπειρία που έχει, ε, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας στις μηχανές. Εγώ δεν ξέρω σε ποια κατηγορία με βάζει ο κύριος Βάντερ Κάμπ. Με βάζει ε, στην αριστερή γραμμή, στη δεξιά γραμμή, στην κεντρό γραμμή, δεν ξέρω. Ελπίζω πάντως όντας στο κέντρο να υποστηρίξει τις τροπολογίες μου. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πώς προσεγγίζουμε τις διάφορες πτυχές. Υποστηρίζω τη γραμμή Van σε σχέση με τα συστήματα πέδησης. Νομίζω ότι είναι πολύ εξισορροπημένη η προσέγγιση για να έχουμε την ε, τον καλύτερο δυνατό αντίκτυπο σε θέματα ασφαλείας. Νομίζω ότι όταν μιλάμε για σκούτερ, για τέτοια δίκυκλα, η προσέγγιση είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τις ε, προαπαιτήσεις ως προς το θέματα βαρύτητας ή ε, σε σχέση με όταν μιλάμε για ποδήλατο. Το θέμα των σκούτερ είναι διαφορετικό ως προς τα δίκυκλα και νομίζω ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα ταχύτητας και υποδύναμης. Νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα πέδησης των σκούτερ και όχι μόνο όταν μιλάμε για ABS και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει βελτίωση κάτω από όλες τις συνθήκες, όχι μόνο όταν υπάρχει επίγουσα ανάγκη. Αυτό δεν είναι ένα σύστημα υποκατάστασης. Ίσως βεβαίως σε επίγουσες καταστάσεις να υπάρχει ένα ειδικό σύστημα πέδησης τύπου ABS. Δεν ξέρω κατά πόσο, κυρία Βέστφαλ, το έχει λάβει υπόψη, αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και την επόμενη εβδομάδα. Τώρα, έμπρακτα, σε σχέση με αυτά που προανέφερα και για τις εκπομπές, δεν αντιτίθεμαι στις βελτιώσεις που προβάλλονται σε σχέση με θέματα απόδοσης των δικύκλων και τρικύκλων αυτών και βεβαίως θα πρέπει να επέλθουν βελτιώσεις, αλλά το βασικό ζήτημα και αυτό θα ήθελα να το θίξω με την Κομισιόν γιατί άκουσα και τους εμπειρογνώμονες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να πω ότι αυτό το σύστημα των Onboard diagnostics ε, μπορεί να επιδέχεται βελτιώσεις, αλλά το θέμα κόστους εκπομπών δεν έχει αναλυθεί επαρκώς. Θα πρέπει να γίνουν ε, ε, βελτιώσεις και στο θέμα κόστους εκπομπών, έτσι ώστε να υπάρχει χαμηλό ε, να υπάρχουν χαμηλές εκπομπές και αυτό πέραν από τις μελέτες κόστους ωφελίας. Από όσο γνωρίζω όμως αυτό δεν έχει συμπεριληφθεί στα δεδομένα της Επιτροπής. Εάν ε, η Επιτροπή με πείσει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε θα, ε, αποσύρω τις τροπολογίες. Τώρα σε σχέση με το σύστημα καυσίμων και τις εκπομπές, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το κόστος είναι σχετικά υψηλό σε σχέση με το συνολικό κόστος των δίκυκλων και αυτό σημαίνει ότι θέλω να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η απόδοση βάση εκπομπών. Δεν λέω ότι θα βελτιώσουμε το σύστημα εκπομπών με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό θα πρέπει να γίνει αναλογικά. Πρόκειται για πολύπλοκες προτάσεις και θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να είμαστε αποδοτικοί και πού δεν είμαστε εκ των πραγμάτων. Τέλος, σε σχέση με τα τετράτροχα ε, ιδιωτικής χρήσης, σας τόνισα ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει λογικά, μέσα στα πλαίσια των ε, τετρακύκλων που μας απασχολούν. Γιατί όταν μιλάμε για ελαφρά οχήματα τα οποία έχουν συγκεκριμένες χρήσεις στον τομέα της γεωργίας, της ε, δασοκομείας και ούτω καθεξής, εδώ μιλάμε για διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα ε, οχήματα επί του οδοστρώματος. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, λειτουργικές απαιτήσεις. Αυτό ελπίζω να είναι ένα θέμα εκκίνησης επί του οποίου θα, συμφωνήσουμε όλοι. Και αν συμφωνήσει και η Επιτροπή, τότε θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να τα συνδυάσουμε και να τα δούμε με βάση την έκθεση Παντζέρη ή την έκθεση Βαντεκάμπ. Στις δικές μου τροπολογίες μιλώ για τεχνικά χαρακτηριστικά σε σχέση με επαγγελματικά γεωργικά οχήματα. Δηλαδή πολλές φορές δεν χρειάζεται να υπάρχουν διαφορικά. Ελπίζω οι συνάδελφοι να συμφωνήσουν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι σημείο εκκίνησης και να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Αυτά ήθελα να πω εγώ ο Σκιώδης. Υπάρχει κάποιος άλλο. Η κυρία Ρούλε. Σας ευχαριστώ. Και εγώ Σκιώδης συγκεκριμένα. Αυτό που κατανόησα από τα όσα είπε ο κ. Βαντεκάμπ είναι ότι δεν θα μας υποβάλει σχέδια συμβιβαστικών τροπολογιών. Βέβαια, δικές μου τροπολογίες είναι αλλιώτικες από τις κυρίες Βέστφαλ. Δεν είπα να βάλουμε τα μοτοποδήλατα στις κατηγορίες των ε, βαριών μοτοσυκλετών. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερο, ιδιαίτερα το ηλεκτρικό ποδήλατο. Εδώ θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να γίνεται η σύγκριση των ε, υποδυνάμεων των ε, οχημάτων αυτών ε, σε σύγκριση μονάχα με ένα τύπο ανθρώπου. Πολύ σύντομα είμαι βεβαία ότι θα έχουμε μεγάλους αριθμούς ηλικιωμένων ανθρώπων, ή σχετικά ηλικιωμένων ανθρώπων, καθώς και αναπήρων, που θα χρησιμοποιούν ηλεκτρικά ποδήλατα. Πρέπει να ανοίξει λοιπόν η αγορά των ηλεκτρονικών ποδηλάτων. Ανεξαρτήτως όμως ε, υποδυνάμεως. Αυτό να εξαρτηθεί δηλαδή από την υποδύναμη αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος. Νομίζω επίσης ότι και οι τρεις και τέσσερις τροχοί σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση δεν επιτρέπει αρκετά περιθώρια διότι αν υποχρεωθούν όλοι αυτοί να υπαχθούν στις κατηγορίες των αυτοκινήτων θα ανοίξει πάρα, θα αναπτυχθεί δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα η αγορά αυτή. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι η οδηγία δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ανάγκες των νέων αυτών αγορών. Ούτε προσφέρει καν μεταβατικές λύσεις και μεταβατικές λύσεις θα με ικανοποιούσαν. Να υπάρχουν κάποιες μεταβατικές λύσεις που να προταθούν στην οδηγία. Εν πάση περιπτώσει αυτό θα χρειαστεί να το συζητήσουμε. Το δεύτερο σημείο που διακρίνεται η άποψή μου από το κ. Βαντεκάμπ είναι ότι υπάρχουν ε, άνθρωποι στη βιομηχανία που λένε ότι ήδη τώρα μπορούμε να μειώσουμε τις εκπομπές και από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να κάνουμε κάθε τι το δυνατόν ώστε οι προσπάθειες αυτές, δηλαδή οι προσφερόμενα, τα προσφερόμενα συστήματα μείωσης των εκπομπών καυσαερίων στην αγορά να είναι ευθυνά. Αντιλαμβάνομαι ότι σε ορισμένα θέματα εκπομπών καυσαερίων Ίσως έχω προχωρήσει πολύ στην διατύπωση της άποψής μου, αλλά νομίζω ότι καλό είναι να σας ασκήσουμε πίεση, γιατί τότε θα, μπορέσετε και θα, θα κινηθείτε και εσείς περισσότερο. Σας ε, συμφωνώ λοιπόν και με το χρονοδιαγραμμά σας και με τα θέματα ABS για, την, ε, για τη διάγνωση με ηλεκτρονικό υπολογιστή του οχήματος. Ε, εκεί νομίζω ότι δεν έχουμε επίσης διαφορές. Άλλος κανείς εκ των σκιωδών. Και συμφωνώ με την κυρία Ρίλε Ρίσεν Παρόδο σχετικά με τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Εσείς κύριε Μάντες. Ε, εγώ θέλω να πω λίγα πράγματα σχετικά με τη διαδικασία. Ο κ. Βαντεκάμπ λέει ότι είναι αδύνατον να υποβάλει συμβαστικέ τροπολογίε. Αυτό είναι κάπως απογοητευτικό. Ίσως να είναι αδύνατον για ορισμένα στοιχεία. Έχω διαβάσει όμω τροπολογίε και βλέπω ότι υπάρχουν κάποια περιθώρια θα μπορούσε να προκύψει ένα καλύτερο αποτέλεσμα με κάποια προσπάθεια. Είμαι βέβαιος ότι ο Βίμ Βαντεκάμ θα θελήσει τελικά να κάνει την προσπάθεια αυτή. Ο πρόεδρος. Νομίζω ότι σε δύο εβδομάδες η συνεδρίαση των σκιωδών στο Στρασβούργο θα είναι αρκετά ε, σκληρή ως διαπραγμάτευση. Ε, τώρα ας ακούσουμε τον κύριο Μαρτίνο που ίσως έχει κάποιες συμβαστικές λύσεις να προτείνει. Uh, σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Βάντερ και τους Σκιώδης. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι διαβάσαμε με μεγάλη προσοχή το προσχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την εργασία. Πολλά θέματα τεχνικής υφής εφήγησαν και έχουμε και πολλές τροπολογίες. Θα ήθελα να σας πω και ήδη είπα ότι χαίρομαι διότι φαίνεται ότι αναλύουμε τις διάφορες επιλογές σε σχέση με το κόστος και την ωφέλεια. Και θα ήθελα να πω ότι ε, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι μπορούμε να καλύψουμε ένα ευρύ φάσμα επιλογών και νομίζω ότι έχουμε καλύψει με το κείμενό μας ε, ως Κομισιόν. Θα ήθελα να αρχίσω με το πιο δύσκολο και διφορούμενο ζήτημα που αφορά τις ε, περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Εδώ είδαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις για την ε, μείωση ή την παράταση του χρόνου, δηλαδή καλύπτουμε θέματα χρονισμού και θα ήθελα να πω ότι έχουμε μία προσέγγιση τριών βημάτων που είναι και ο σωστός συμβιβασμός. Τελικός στόχος είναι να μην έχουμε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων που να επιδεινώνουν την όλη κατάσταση και το περιβάλλον. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι συνολικές εκπομπές στο οδόστρωμα, οι οποίες να μην αυξάνονται αλλά να μειώνονται. Η τρίπτυχη αυτή προσέγγιση, η προσέγγιση τριών βημάτων, θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή και αποτελεί τη βέλτιστη δυνατή λύση. Τα άλλα συσχετιζόμενα στοιχεία που θίξατε εσείς πρόεδρε και ο εισηγητής σε σχέση με τα on-board diagnostics, αυτό το θέμα δεν μας απασχόλησε στη μελέτη. Είχαμε και τις υποδείξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν αρκετές ελλείψεις, όπως μας είπαν οι εμπειρογνώμονες. Θα ήθελα όμως να πω ότι η δική μας προσέγγιση καλύπτει βασικές απαιτήσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και να ακολουθήσουμε όλους τους κατασκευαστές των διαφόρων κατηγοριών προϊόντων. Ξέρετε ότι αρχίζουμε με την ε, υποχρέωση που αρχίζει από το 2017 για τα MOPID και τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Ε, για τα ηλεκτρικά ποδήλατα αυτό το πλαίσιο θα ισχύσει από το 2021. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρξει μία ε, υποστήριξη σε σχέση με τα ηλεκτρικά οχήματα τα οποία αποκλείονται από τις ε, περιβαλλοντικές προδιαγραφές μέσα στα πλαίσια των κατοφλίων on-board diagnostics. Το άλλο ζήτημα αφορά την διάρκεια των εκπομπών και την ε, ε, πτητικότητά τους. Αυτό που μας ενδιαφέρει και εδώ θα ήθελα να τονίσω του στόχου μας, είναι ότι θα πρέπει να γίνουν δοκιμές συνέχειας ή διάρκειας και να μην είναι μόνο μια άσκηση επιχάρτου χωρίς να υπάρχουν βελτιώσεις στον τομέα αυτό. Θα θέλαμε να δούμε τι πρόοδος έχει επιτελεστεί για να ε, ε, επαναορίσουμε τις δοκιμές αυτές. Από όσο γνωρίζω, στις υπάρχει μία περιφερειακή προσέγγιση, αποκεντρωμένη προσέγγιση, ιδιαίτερα σε σχέση με τα οχήματα κατηγορίας 4. γιατί είναι διαφορετική κατάσταση ανάλογα με το προϊόν για το οποίο μιλάμε. Η κατάσταση διαφέρει μεταξύ Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, και ΕΠΑ σε σχέση με τα MOPID. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ένα σύστημα επέδυσης για τα οχήματα αυτά Προσπαθήσαμε να φτάσουμε σε μια ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας και κόστους, καθώς και στόχου υψηλής ασφαλείας. Ως προς ε, μέτρα αντιστάθμισης, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προβούμε σε μία ανάλυση κόστους ωφελίας έτσι ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Το άλλο στοιχείο, τα άλλα δύο στοιχεία είναι αυτά τα οποία προανέφερα, δηλαδή η εμβέλεια και η υποκατηγοριοποίηση καθώς και τα ηλεκτρικά δίκυκλα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε παραμέτρους. Εδώ ως Επιτροπή θα θέλαμε να τονίσουμε ότι έχει μεγάλη σημασία να ε, προβάλλουμε και επιπρόσθετες παραμέτρους, να λάβουμε υπόψη την ταχύτητα καθώς και την υποδύναμη σαν βασικές παραμέτρους. Διότι υπάρχει άλληλος συσχετισμός μεταξύ ταχύτητας και υποδύναμης, καθώς και ταχύτητας και ασφάλειας. Εδώ μιλώ για τη διαφορική ταχύτητα μεταξύ ε, ενός οχήματος και ενός άλλου. Άρα και για τα δίκυκλα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διαφορική ταχύτητα μεταξύ δικύκλου και πεζού. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν ε, και αυτές τις δύο παραμέτρους, δηλαδή την ταχύτητα και την υποδύναμη. Ε, ζητώ συγγνώμη αν καταχράστηκα του χρόνου σας, αλλά νομίζω ότι κάλυψα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ανέφερε ο εισηγητής και η Σκιώδης. Αν ξέχασα κάτι να μου το υπενθυμίσετε ή αν θέλετε επιπρόσθετες δραστηριότητες ως προς τα ATV. Τα οχήματα παντός εδάφους προσπαθούμε να καλύψουμε διάφορες κατηγορίες και μπορούμε να δεχτούμε βελτιώσεις, αλλά ένα από τα στοιχεία που αναφέρατε, τα στοιχεία που αναφέρατε, που αναφέρατε εσείς είναι απόλυτα λογικά. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Ε, η ανταλλαγή απόψεων ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη, αλλά οι σκιώδεις θα συνεργαστούν με τον εισηγητή τις επόμενες εβδομάδες μέχρι την ψηφοφορία. Στο τέλο μπορεί να μην συμφωνήσουμε με όλα τα στοιχεία επιτόπιτο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Κύριε αν θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ μερικά λεπτά κύριε Πρόεδρε, αν συμφωνείτε. Κυρία Στήλε έφυγε. Αλλά θα έρθω σε επαφή με την κυρία Βέστφαλ. για τα σχόλια της ε, για τα ABS και τα CBS. Η κυρία Ριούλε είπε ότι η κυρία Βεστφάλ δεν διατίθεται να συμβιβαστεί. Αν μου επιτρέπετε να εκφραστώ ούτως. Και εγώ δεν ξέρω αν μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις επιθυμίες της. Στην παρατήρηση του κυρίου Μάντερς. Εμείς σήμερα μιλάμε για έναν τεχνικό κανονισμό. Μιλάμε για τα δίτροχα οχήματα από τεχνικής πλευράς. Όταν μιλάμε όμως για τεχνική δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ασφάλεια. Πρόκειται, είπαμε, για τεχνικού χαρακτήρα κανονισμό. Εγώ δεν κάνω καμία διάκριση βέβαια σε αυτό διότι και για μένα η ασφάλεια του οδηγού είναι το κυρίαρχο και το πιο ουσιαστικό, αλλά θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή όχι. Για τις παρατηρήσεις σας είναι σαφέστατες, για τις εκπομπές. αλλά δεν μιλήσατε για τα τεστ διάρκειας. Ε, είστε ο μόνος που καταθέσατε μία τέτοια τροπολογία. Θα μπορούσατε λοιπόν να ξαναδείτε την τροπολογία σας. Παρατήρηση της κυρίας Ρούλε. Μα δεν υπάρχει παρεξήγηση για το ΣΕΜΠΕΣ και το ΑΕΜΠΕΣ μεταξύ μας. αλλά ο πιο ισχυρός κινητήρας Οποιοςδήποτε μάλλον ισχυρότερος κινητήρας μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ποδήλατο. Πρέπει να φανταστούμε εμείς μέχρι ποια όρια μηχανής μπορούμε να βάλουμε στο ποδήλατο. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ας πούμε, να οδηγεί ένα ηλεκτρικό ποδήλατο 60 χιλιόμετρα την ώρα και να μην φοράει κράνος. Και αν κάποιος οδηγεί ένα μοτοποδήλατο 25, με 25 χιλιόμετρα την ώρα, ε, και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η αγορά των ηλεκτρικών ποδηλάτων είναι μια τεράστια αγορά. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη για τις εκπομπές. Οι πράσινοι θέλουν να προχωρήσουν μακρύτερα. Εσείς θέλετε να προχωρήσουμε πιο αργά. Ας επιλέξουμε λοιπόν τη μέση λύση του Βαντερκάντ. Τώρα πάντοτε προσεγγίσαμε συμβιβαστικές τροπολογίες αυτό το κοινοβούλιο παρότι λέγεται το αντίθετο. Εγώ τι να κάνω, τι θέλετε να κάνω, να κλέψω ένα κείμενο της Κομισιόν, να το κάνω και αυτό άμα αυτό ικανοποιήσει τον κύριο Μάντερς. Είμαστε σε μια φάση εναρμόνισης και πρέπει να είμαστε ειλικτρινείς με τους δε. Είμαι έτοιμος να υποβάλω τροπολογίες ε, για το κείμενό μου, αλλά για το κείμενο της Κομισιόν δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν με πληρώνουν γι' αυτό. Ευχαριστώ. Έχουμε πολλή εργασία μπροστά μας, η οποία θα γίνει πριν από τις ε, ψηφοφορίες. Εγώ δέχομαι τα δεδομένα που μας προαναφέρατε. Υπό την αιγίδα σας λοιπόν θα προχωρήσουμε. Τώρα θα μας απασχολήσει το επόμενο θέμα που, αφορούν, που αφορά τις τροπολογίες της έκθεσης Hansling σε σχέση με τις 58 δηλαδή τροπολογίες της διαδικασίας αμοιβαία αξιολόγησης της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Ο κύριος Μάντερς είναι εδώ, εγώ είμαι εδώ, Σκιώδης. Η κυρία Γκέπχαρτ δεν είναι εδώ και δεν υπάρχει κάποιος από τους πρασίνους. Ούτε ο κύριος Τριανταφυλλίδης είναι παρόν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα απαντήσει κάποιος από τους σοσιαλιστές, αλλά θα ήταν σκόπιμο να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια για να μας μιλήσει για τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στην έκθεσή της. έχω. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ όλους για τις τροπολογίες που υποβάλατε σε σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης. Έχετε προβάλει 58 τροπολογίες και κατά την άποψή μου αυτό δείχνει ότι εμπολής υποστηρίζεται την ε, γνωμοδότησή μου προσπαθήσατε να διευκρινίσετε ζητήματα που δεν καλύπτω εγώ και αφορούν τρία βασικά ζητήματα. Καταρχήν, την ε, πρώτη μας εμπειρία σε σχέση με την αμοιβαία διαδικασία αξιολόγησης οδηγίας για τις υπηρεσίες, τη μελλοντική χρήση της αξιολόγησης και τα αποτελέσματα των, της μελλοντικής δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς εξαιτίας, μάλλον με βάση και χάριν αυτής της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης. Θα ήθελα να τονίσω ότι πολλές από τις τροπολογίες θα τις υποστηρίξω καθώς και η πολιτική μου ομάδα στο εγγύς μέλλον. Όταν ε, δούμε πώς θα ε, γνωμοδοτήσουν οι διάφορες επιτροπές. Θα ήθελα να σας υποβάλω δηλαδή τροπολογίες συμβιβασμού εκεί όπου θα μπορέσω. Ασχοληθήκαμε με αυτές, ε, όλες αυτές τις πτυχές τόσες φορές που θα θέλαμε η οδηγία περί υπηρεσιών να μπορεί να εφαρμοστεί από τους επιχειρηματίες και να είναι και ιδιαίτερα επικοδομητική για τις υπηρεσίες. Στο άρθρο 15 αναφερθήκατε στην οδηγία σε όλες τις, τις εκφάνσεις και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο αυτή η οδηγία έχει εφαρμοστεί και κατά πόσο επηρεάζει την κατάσταση των υπηρεσιών. Προβλέπουμε τη δημοσίευση αυτής της ανάλυσης κατά το τέλος του έτους. Σύμφωνα με το άρθρο 41 της ε, Οδηγίας Υπηρεσιών, η Επιτροπή θα πρέπει να μας υποβάλει μία έκθεση για την εφαρμογή της Οδηγίας Υπηρεσιών. και ελπίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ε, θετικές αποτιμήσεις, σε μια θετική αποτίμηση στο μέλλον. Ο κύριος Χάρμπορ στην τροπολογία 29 μιλάει για διαφάνεια, μεθοδολογία, αποσαφήνιση και ε, το γεγονός θα πρέπει να βασιστούμε στη μέθοδο εφαρμογής. Θα ήθελα οι εκπρόσωποι της Επιτροπής να μας μιλήσουν για αυτή τη μέθοδο εφαρμογής ή δυνατόν ακόμα και σήμερα. Ως προς ε, άλλες τροπολογίες που δεν μπορώ να υποστηρίξω, εδώ υπόκειται και η τροπολογία 32, η 34 επίσης, Κάνφιν και Χάρμπορ, που δεν σχετίζεται με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Γι' αυτό νομίζω Και νομίζω ότι αυτά δεν θα πρέπει να μας ζητήματα, τέτοια ζητήματα δεν θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Ως προς τροπολογία 34, ως και ως προς τη χώρα προέλευσης, το θέμα αυτό είχε ήδη λήξει το 2009, όταν εγκρίναμε την οδηγία. Και δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη λύση. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τις διασυνοριακές υπηρεσίες. Νομίζω, νομίζω ότι η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης μας δίνει μία επίκαιρη εικόνα για το πώς έχουν ε, ε, δράσει τα κράτη-μέλη σε σχέση με την κατάσταση μέχρι τούδε. Όμως δεν έχουμε μία συνολική εικόνα, γιατί δεν περιλαμβάνονται μερικά κράτη-μέλη. Σε ορισμένες τροπολογίες αναφερθήκατε σε θέματα υπηρεσιών, πόσο σημαντικές είναι οι υπηρεσίες για τις οικονομίες μας, με νέες θέσεις εργασίας, με την αναπτυξιακή πορεία των οικονομιών μας ε, μέσα στα πλαίσια της κρίσης της υπάρχουσας και άλλων υποφαινομένων κρίσεων. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τούδε και να απαιτήσουμε και άλλες εξελίξεις. Το Δεκέμβριο θα διανύουμε τα δύο χρόνια μετά από την έγκριση της οδηγίας, γι' αυτό θα πρέπει να γίνει ένας απολογισμός. Πιστεύω ότι η έκθεσή μου καθώς και οι τροπολογίες σας θα δώσουν μια νέα όθηση στις συζητήσεις για την οδηγία περί υπηρεσιών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η οδηγία περί υπηρεσιών είναι ένα από τα βασικότερα νομικά κύματα τα οποία έχουν προπαρασκευαστεί και εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Τώρα θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας γνωμοδοτήσεις, να μου πείτε τι σκέφτεστε ως σκιώδης και ιδιαίτερα εσείς κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κυρία Χάνσλικ για την σαφή σας ανάλυση. Η κυρία Γκέπχαρτ δεν είναι παρούσα. Ποιος θα μιλήσει από τους σοσιαλιστές. Εσείς κύριε Μάντερς. Βεβαίως. Πολύ ευχαριστώ, πολύ ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Αυτή τη η προσέγγιση είναι πάρα πολύ χρήσιμη για την βελτίωση της οδηγίας για τις υπηρεσίες και τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης που μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές οδηγίες, όχι μόνο στην οδηγία για τις υπηρεσίες παρακολούθηση της εσωτερικής αγοράς για παράδειγμα. Οι οδηγίες εφαρμόζονται διαφορετικά από τη μία χώρα στην άλλη, οπότε η εσωτερική αγορά και αυτή δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Το αποτέλεσμα αυτής της αμοιβαίας αξιολόγησης θα καταδείξει ότι τα κράτη-μέλη βρίσκονται ακόμη σε φάση ανταγωνισμού και δεν βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν παράγοντα ενοποίησης ε, και παράγοντα γενικής πρόοδου. Άμα βλέπουμε λοιπόν εμείς με στραβό μάτι το γείτονα με προστατευτικές ε, διαθέσεις, ε, αυτό στρέφεται πλέον σε, μια δεύτερη φάση εναντίον των ιδίων των κρατών μελών. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο στοχεύει στη βελτίωση της εσωτερικής αγοράς και της συνεργασίας. Ευχαριστώ την εισηγήτρια που υποστήριξε τις τροπολογίες μου και εγώ υποστηρίζω τη δική της άποψη. Βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Θέλουμε να βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά. Και ελπίζω ότι μπορούμε να φανταστούμε και άλλες δυνατότητες. Άμα φανεί δηλαδή μετά από αυτήν την ανάλυση ότι ορισμένα κράτη καταχρώνται της ερμηνευτικής τους δυνατότητας, τότε μπορούμε να λάβουμε μέτρα και να δράσουμε εναντίον αυτών των κρατών μελών. Κυρία Ρίουλε, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, όχι. Θα ήθελα να σχολιάσω, Ναι. Χαίρομαι. Κυρία Χάντσλικ, που θεωρείτε ότι οι τροπολογίες μου προσθέτουν στην έκθεσή σας. Από τη δική μου πλευρά το αποτέλεσμα της, του μείγματος της αξιολόγησης σε τομείς προτεραιότητας για την βελτίωση της διαμεθοριακής οικονομικής ε, ανάπτυξης νομίζω ότι είναι σημαντικά. Έχετε όλα αυτά τα δεδομένα επιτάπητος και αναμένουμε να τα χρησιμοποιήσετε ώστε να καθορίσετε κάποιες προτεραιότητες σχετικά με το πού θα πρέπει να ασκηθεί πίεση από πλευρά χωρών μελών να ανοίξουν οι αγορές ώστε να δημιουργηθεί απασχόληση και δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε όντως αυτόν τον οικονομικό δυναμισμό, απεγνωσμένα τον χρειαζόμαστε και τη δημιουργία απασχόλησης και μάλιστα δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο σε αυτή την αξιολόγηση. Το σημαντικό είναι επίσης ότι πρόκειται πληροφορίε που χορηγούν οι ίδιες οι χώρε μέλη. Δηλαδή δεν, έρχονται, δεν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει άνωθεν πράγματα στις χώρε μέλη. Και αυτό είναι ιδιαίτερα αξιόλογο για την εφαρμογή της οδηγία τη ενέργεια αγορά. Εάν η Επιτροπή μας υποστηρίξει, θα είναι σαφές το μήνυμα που δίνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα όσα προωθείτε για την διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης. Ευχαριστώ λοιπόν που στηρίζετε τις τροπολογίες μου. Θα έπρεπε να είχα καλωσορίσει τον κύριο Μάρτιν Φρέν προηγουμένως που είναι τώρα αρμόδιος για την εφαρμογή της οδηγίας υπηρεσιών. Με την άδειά σας κύριε θα τον παρακαλέσω να σχολιάσει τις τροπολογίες και μετά θα δώσω το λόγο σε εσά για να μας πείτε πώς θα προχωρήσετε και αν θα υποβάλλετε συμβαστικές τροπολογίες. Μάρτιν Φρέν. Ευχαριστώ και εσάς και την εισηγήτρια καθώς και τους Σιώδης συμφωνούμε απολύτως με την ανάλυση της κυρίας Χάντσικ. Πολλές από τις τροπολογίες όντως βελτιώνουν την πρότασή μας. Άκουσα το μήνυμά σας, το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Λίγα λόγια για την μελέτη ε, οικονομικών επιπτώσεων και τον εντοπισμό ορισμένων προτεραιοτήτων όπως ε, εξηγήσαμε και στον ανακοινωθέν μας την ανάλυση αυτή, τη μελέτη αυτή θα την κάνει η αρμόδια γενική διεύθυνση στη βάση μελετών που προσπαθούν να προβλέψουν την οικονομική, τις οικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής της οδηγίας στη βάση των πληροφοριών που μας έχουν χορηγήσει οι χώρες μέλη και από άλλες πηγές. Δεν θα είναι πλήρης η απεικόνηση των αποτελεσμάτων της ε, οδηγίας η οποία είναι εξαιρετικά νεαρά ακόμη και δεν έχουμε όλες τι πληροφορίες. Αλλά θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά στα οικονομικά δεδομένα, στις μελέτες που έχουμε ε, συντάξει και στη βάση των προτάσεων που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προετών ακόμη. Αυτά θα βασιστούν στη μεθοδολογία που είχε χρησιμοποιηθεί τότε από τα διάφορα οικονομικά ε, ιδρύματα, καλά βέβαια πάντοτε με την απαραίτητη επιστημονική ε, θεμελίωση ο ίδιος δεν είμαι επιστήμονας, ειδικός επιστήμονας, δεν θα μπορέσω να σας αναπτύξω τις λεπτομέρειες της μεθοδολογίας, αλλά θα το πράξουμε αυτό στο μέλλον. Γιατί οι συνάδελφοι μου της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να σας τα εξηγήσουν. Ορισμένες τροπολογίες δικές σας κύριε Χάρμπορ σχετικά με την διαφάνεια που θα πρέπει να εξασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν συζητεί με τι χώρε μέλη, καθώ επίση ο εντοπισμό των προτεραιοτήτων. Εμεί ασφαλώ θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διαφανής. όπως άλλωστε έχει συμφωνηθεί με πρωτοβουλία της Επιτροπής της μεταξύ των θεσμικών οργάνων για την διαφάνεια που έχει αποφασιστεί καθώς και για τις δοκιμασίες απόδοσης, performance checks και αυτά θα μπορέσουν να τα εξετάσουν οι συναδελφοί σας στην ιστοσελίδα μας και να δουν ότι συζητούμε με τις χώρες μέλη τα θέματα αυτά, καθώς επίσης και με ποιο τρόπο θα προχωρήσουμε. Θα σας δείξει αυτό ότι συμφωνούμε απολύτως με το πνεύμα διαφάνειας που ζητεί ο κ. Χάρμπορ στις ε, τροπολογίες του. Νομίζω ότι μπορώ να αρκεστώ σε αυτά τα λίγα σχόλια. Βεβαίω υπάρχουν ορισμένε τροπολογίε που θεωρούμε ότι δεν μα βοηθούν τόσο πολύ. Κυρίω για θέματα που ασφαλώ είναι σημαντικά, αλλά που ίσω να μην έχουν τόσο άμεση διασύνδεση με τα θέματα που συζητούμε τη μελλοντική αξιολόγηση, δηλαδή, ίσως μάλιστα ούτε και εξετάζοντας και ε, συζητήσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, καθώς και για την μελέτη οικονομικού χαρακτήρα που προαναγγείλατε. Βρίσκω ότι έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά. Τώρα η κυρία Χαντσλίκ μπορείτε αν θέλετε να απαντήσετε και στην Κομισιόν αλλά και στους Κιώδης και να μας αναπτύξετε και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμά σας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, μελέτη οικονομικού αντικτύπου. Νομίζω ότι το έγγραφο αυτό μας δείχνει ότι η οδηγία περί υπηρεσιών έχει μεγάλη σημασία για την διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Αναμένουμε αυτό το έγγραφο για το τέλος του έτους. Όπως σας είπα πριν, μπορώ να συμφωνήσω με αρκετά αρκετές ε, τροπολογίες σας, διότι εμπλουτίσουν το εγγραφό μου και αποτελούν προσθέμενη αξία. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τις αναλύσω και ευχαριστώ τον Πρόεδρο και για, για τις τροπολογίες του. Και οι περισσότερες θα έχουν ένα που σημαίνει ότι θα τις υποστηρίξω. Θα ψηφίσουμε στο εγγύς μέλλον. Γι' αυτό αυτό την επόμενη εβδομάδα θα δώσω στους σκιώδεις τις τροπολογίες συμβιβασμού και εάν θέλετε μπορούμε να συναντηθούμε και να συζητήσουμε τους συμβιβασμούς πριν από την επόμενη συνάντηση, γιατί την επόμενη φορά θα πρέπει να ψηφίσουμε για το έγγραφο αυτό στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για τις τροπολογίες σας και νομίζω ότι η διαδικασία αυτή αμοιβαία αξιολόγησης είναι κάτι που χρειάζεται άμεσα. Thank you Ευχαριστούμε πολύ. Αναμένουμε τις εργασίες σας μέχρι την ψηφοφορία στις 19 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε και την Επιτροπή. Προτρέχουμε κάπως για μία φορά. Βλέπω ότι ο κύριος Κρόιτσμεν είναι εδώ. Ελπίζω να είναι όλοι, ιδιαίτερα η ομάδα της Επιτροπής. Πριν αρχίσουμε, θέλετε να διακόψουμε για πέντε λεπτά. Ας διακόψουμε για πέντε λεπτά. Και θα συνεχίσουμε λίγο πριν ε, τις πέντε, έτσι ώστε όλοι να είναι παρόντες. So Διακόπτουμε για πέντε λεπτά. Πέντε, επτά λεπτά για να είναι όλοι παρόντες για να απαντήσουν στον κύριο Κρόιτσμαν.

ladies and gentlemen, I think we're ready to resume. I hope everybody's here. Ελπίζω όλοι να είναι παρόντες. Ξαναρχίζουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Ελπίζω όλοι να είναι παρόντες ως προς την ε, άκρος ενδιαφέρουσα και σημαντική έκθεση του κύριου Κρόιτσμαν Ε, συζητώ με τον συνάδελφο για τις τροπολογίες του. Δεν ήμουν και ιδιαίτερα ευτυχής και προσπάθησα να τον επιράσω. Προσπάθησα να τον πείσω, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Θα... Ο, να κάνω μια εισαγωγή πριν αρχίσετε. Και ιδιαίτερα για το κοινό μας, το οποίο μας παρακολουθεί από το διαδίκτυο. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι τώρα θα ασχοληθούμε με την έκθεση Κρόιτσμαν. Πρόκειται για μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σύνδεση στην εσωτερική αγορά. Νομίζω ότι είχαμε 271 τροπολογίες, αν δεν κάνω λάθος. Μετά θα δώσω το λόγο στους κοιόδης. Ο κύρος Άμπατ θα έρθει λίγο αργότερα Σαλτεμόζερ είναι παρόν, η κυρία Ρούλε εδώ, εδώ. Φόξ εδώ, Σαβίνη, Απόν και έχουμε την κυρία Μπρόντε από την ε, Επιτροπή η οποία θα μας απαντήσει. Ωραία. Σας καλωσορίζουμε και σε εσάς. Η κυρία Μπρόντε θα μας ε, μιλήσει για την άποψη της Κομισιόν Άρα ο κύριος Κρόιτσμαν θα λάβει το λόγο και μετά θα μας μιλήσει για το πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε έναν εύλογο συμβιβασμό. Κύριε Κρόιτσμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Έχουμε πράγματι 271 τροπολογίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώτης και όλους όσους υπέβαλαν τροπολογίες. Γιατί οι περισσότερες τροπολογίες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή με υποστήριζουν. Α, ο κύριος De μόλις μπαίνει. Οι τροπολογίες του κινούνται προς διαφορετική κατεύθυνση. Θα επανέλθω αργότερα δεν θα ήθελα να, να σταθώ στη δεξιά ή την αριστερά, όπως είπε ο κύριος Βάντερ Κάμπ. Θέλουμε να φτάσουμε σε ένα σύστημα ευρωπαϊκής εμβέλειας. Ο κύριος Σαλτεμόζερ ίσως ε, θα ήθελε να αφήσει τα πράγματα ως έχουν. Και ο κύριος Γκρέκ θέλει να έχουμε ένα ανοιχτό σύστημα. Ο κύριος Φόξ θα ήθελε να υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα και πολλοί τάσσονται υπέρ του status quo. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μία λύση μεταξύ όλων αυτών. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε καλώς. Βασιζόμαστε στην ιδέα ότι θα πρέπει να έχουμε μία εξισορροπημένη προσέγγιση. Γι' αυτό έχω υποβάλει και προτάσεις συμβιβασμού, τις οποίες θα συζητήσουμε θα σας δώσω ένα κατάλογο συστάσεων για να έχετε μία σαφή ιδέα και να δούμε σε τι συμβιβασμούς μπορούμε να φτάσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε βελτιώσεις. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Βεβαίως έχει βελτιωθεί η έκθεση εγώ δεν είμαι υπέρ των εθνικών μονοπωλίων, αλλά δέχομαι ότι ορισμένα κράτη-μέλη θα ήθελαν να περιορίσουν αυτά τα τυχερά παιχνίδια online και θα ήθελαν να υπάρχει προστασία του καταναλωτή να καταπολεμηθεί και η εγκληματικότητα και θα πρέπει να γνωρίσουν οι καταναλωτές, οι καταναλωτές ότι υπάρχει διαφάνεια και δεν υπάρχουν διακρίσεις. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης των αδειών του συστήματος αδειοδότησης και το διοικητικό κόστος θα πρέπει να συρρυκνωθεί. Αυτό βεβαίως δεν αποκλεί περαιτέρω εθνικούς διακανονισμούς ή κανονισμούς γενικότερα, και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την απάτη και να προωθήσουμε την προστασία των νέων. Χρειαζόμαστε ελάχιστες προδιαγραφές. Αυτό δεν σημαίνει ε, χαμηλά κατόφλια, αντίθετα σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους να έχουν πιο αυστηρούς κανόνες σε σχέση με τους κανόνες που προανέφερα ελπίζω να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις έγνοιες του κυρίου Σάλτεμοζε. Ε, αν δεν φτάσουμε σε μια συμφωνία, τότε η Επιτροπή θα πρέπει να εισαγάγει ελάχιστες προδιαγραφές. Θα ήθελα δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μια ευρεία βάση εργασίας για αυτή την έκθεση, έτσι ώστε να πιστεί η Επιτροπή να κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Και οι περισσότεροι συνάδελφοι συμφωνούν με αυτή την προσέγγιση και συμφωνώ με τον συνάδελφο που ε, είπε προηγουμένως ότι κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να ορίσει μία αρχή η οποία θα συνεργαστεί με το ευρωπαϊκό επίπεδο για να θεσπιστούν κανόνες για, την, ε, για τα τυχερά παιχνίδια. Και αυτά θα πρέπει να βασιστούν σε εφιστάμενες ε, δομές. Χρειάζεται επίσης και ένας κοινός ορισμός για την απάτη στα τυχερά παιχνίδια, καθώς επίσης η ποινική δίωξή τους, των απατών αυτών δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της ακαιρεότητας στα τυχερά παιχνίδια. Και για να ωφεληθούν κυρίως ε, τα, ο ερασιτεχνικός αθλητισμός όπου επίσης πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά των καταχρήσεων. Ο κ. Σφάπ και άλλοι ζήτησαν την επιβολή του γαλλικού προτύπου όταν μιλούμε για χρηματοδότηση ωστόσο αθλητικών, ε, αθλητισμών, παιδιών κτλ. Αρχικά εγώ δεν είχα κάνει σχετικά προτάσεις γιατί όλα αυτά θεωρώ ότι καλύπτονται από την αρχή της επικουρικότητας το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά που προκύπτουν από τα έσοδα από την έγκριση αδειών, από τη χορήγηση αδειών, θα πρέπει να είναι υπόθεση των χωρών μελών. Βεβαίως, αν υπάρχουν άλλες απόψεις, είμαι ανοιχτό στο θέμα αυτό. Μπορεί όμως να θεωρηθεί, όπως είπα πριν, ότι καλύπτεται η υπόθεση από την αρχή της επικουρικότητας. Αν θα τα κρίνουν οι χώρες μέλη. Ο Δόκτωρ Σφάπ έχει δίκιο ότι και νόμιμα τα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να λειτουργήσουν χωρίς κάποιο βαθμό διαφήμισης. Αλλά πρέπει να ρυθμιστούν τα θέματα αυτά και για την καταπολέμηση της μαύρης αγοράς. Με κοινέ προδιαγραφές. Το ίδιο για τους χορηγούς, sponsors. Και κυρίως με γνώμονα την προστασία του καταναλωτού. Εγώ σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον ρώτησα πώς τα έχουν ρυθμίσει εκεί. Μου είπαν ότι οι ε, σύνδεσμοι αθλητικών συλλόγων δεν θέλουν ε, στοιχήματα για ποδόσφαιρο, για φούτμπολ δηλαδή, μπάσκετμπολ κλπ. Αν θέλαμε και εμείς να το κάνουμε εδώ, αλλά κανείς δεν το θέλει, θα έλυγε το πρόβλημα γιατί δεν θα επιτρέπονταν τότε στοιχήματα για ποδοσφαιρικούς αγώνες. Και υπάρχει και κάτι άλλο εκεί και εκεί ο κύριος De έχει κάνει μια μοναδική τροπολογία που θεωρώ ότι πρέπει να συζητηθεί. Οι Αμερικανοί απαγορεύουν να έχουν οι ενδιαφερόμενοι πιστοτικές κάρτες για να παίζουν επιγραμμικά, online gambling δηλαδή. Πιστοτικές κάρτες και ε, λογαριασμούς πιστοτικών καρτών για παράνομους προσφέροντες. Εκεί πρέπει να απαγορευτούν αυτά. Για μας το λέω αυτό εδώ. Εφόσον πρόκειται για παράνομες δράσεις, αν το κάνουμε αυτό, έχουμε χτυπήσει το παράνομο αυτό εμπόριο. Και εδώ νομίζω συμφωνούν όλοι. Εγώ θα το συζητήσω με τους ε, σκιώδεις συγητές. Η ιδέα αυτή μου ήρθε όταν διάβασα την τροπολογία σας κύριε συνάδελφε. Εσείς δεν θέλετε βέβαια να ρυθμιστεί τίποτα λέτε. Αυτό δεν έχει νόημα γιατί θέλουμε βεβαίω να τηρηθεί η αρχή τη επικουρικότητα. Μην κάνουμε όμω τίποτε όπω προτείνετε εσεί. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν εσφαλμένο δρόμο. Γιατί θα διατηρηθούν τα μονοπόλια, τα κρατικά μονοπόλια που διαθέτουν ορισμένε χώρε. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η παρούσα κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Ως επόμενο βήμα θα προχωρήσω στις 16 Ενάτου σε διαβούλευση με τους κοιόδης με ψηφοφορία στην Ολομέλεια να προβλέπεται περί τα τέλη Οκτωβρίου. Έλαβα 71 τροπολογίες, όλες σχεδόν κατευθύνονται στην ίδια κατεύθυνση, ότι πρέπει κάτι να γίνει δηλαδή, στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αν θα καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε και τους Βρετανούς που θέλουν να ανοιχθεί ακόμα περισσότερο η αγορά, αυτό δεν ξέρω αν θα το επιτύχουμε. Σας ευχαριστώ πάντως που με παρακολουθήσατε. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Η προσέγγιση σας είναι αξιέπαινη. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι θα μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της ε, εκθέσεως πρωτοβουλίας με τον τρόπο αυτό, γιατί θα δώσουμε έτσι μια κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω θα το επιτύχουμε χάρη στις προσπάθειές σας. Υπάρχουν βέβαια οι φιλελεύθερες απόψεις ορισμένων συναδέλφων μας, αλλά και πιο συντηρητικές από άλλες πλευρές του σώματος. Πάντως, εσείς ασφαλώς μπορείτε να τις γεφυρώσετε, τις όποιες διαφορές υπάρχουν μεταξύ φιλελευθέρων και συντηρητικών. Ο κ. Αμπάντη είναι παρόν. Θέλετε να μιλήσετε τώρα και δεν ήσασταν όμως από την αρχή ή προτιμάτε να περιμένετε να μιλήσετε στο τέλος. Μάλιστα, στο τέλος, καλά. Θα σας δώσω το λόγο λίγο αργότερα. Ο κ ο κ. Φόξ, επίσης και Ρίλε, ο κ. Ντιόν και ο κ. Σαμπάντ. Έχουμε και τον καθηγητή Δεκάμπος. Επιθυμεί κανείς άλλος να ομιλήσει. Έχουμε χρόνο. Στο τέλος θα δώσω τον λόγο στον κύριο Κούντσμαν να δούμε αν έχει ε, πλησιάσει κάπως το όραμά του ε, για ένα πακέτο δηλαδή συμβασμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια σειρά τροπολογιών. Είναι συνολικά 271 και αυτός ο μεγάλος αριθμός δείχνει το έντονο ενδιαφέρον των ε, συναδέλφων καθώς επίσης και το γεγονός ότι υπάρχουν μεγάλες εθνικές διαφορές στις ρυθμίσεις για τα τυχερά παιχνίδια. Και η έκθεσή μας πρέπει να το αποδίδει αυτό. Συμφωνώ πάντως με την έκθεση του κ. Κρότσμαν που λέει ότι μπορεί να, είναι, να γίνει τελικά εξαιρετική η έκθεση αυτή. Συμφωνώ και θεωρώ ότι χρειάζεται να γίνουν κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Είπε προηγουμένως ο κ. Κρότσμαν ότι ο κ. Κρέκ και εγώ, από την ομάδα μου ο ίδιος δηλαδή, ε, βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Σωστό. Υπάρχουν διαφορές απόψεων και νομίζω λίγο πολύ σε όλες τις ε, πολιτικές ομάδες. Τουλάχιστον στο Λαϊκό Κόμμα υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Εγώ δεν είμαι αρνητική στην προσπάθεια να ξεύρουμε κάποιες λύσεις. Θα ήθελα να βρεθεί κάποια λύση στο ευρωπαϊκό επίπεδο για ε, τα τυχερά παιχνίδια. Απλώς είμαι επιφυλακτική για το αν θα πρέπει να λάβει τη μορφή οδηγία. Θα ήθελα να δω να συνεργάζονται περισσότερο οι αρχές των χωρών μελών. Και νομίζω ότι υπάρχουν κατάλληλε προτάσει που περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών των τροπολογιών. Η προσέγγιση του κ. Αμπάντ, για παράδειγμα, Πάντως, τα όσα είπαν οι κύριοι Μπούσετιλ, Φόξ και Φιέλνερ, είναι μια προσέγγιση που δεν υποστηρίζω απαραίτητα. Η προσέγγιση που δεν μου αρέσει είναι να ανοιχτεί μια μεγάλη ενιαία αγορά για τα τυχερά παιχνίδια. το τυχερό παιχνίδι είναι οικονομική δραστηριότητα, αλλά ε, με όλο ιδιαίτερο χαρακτήρα και εκεί απαιτούνται ιδιαίτεροι κανόνες. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι είναι μια συνήθι οικονομική δραστηριότητα. Αναμένω λοιπόν την περαιτέρω συνεργασία και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα στηριχθεί σε μεγάλη πλειοψηφία από τα μέλη της ε, Επιτροπής μας. Ευχαριστώ κύριε Σαλεμόζε. Ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κρότσμαν για την εργασία του. Συμφωνώ με τους στόχους του ότι χρειαζόμαστε μια ευρεία προσέγγιση για να αναγκάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί, διότι το χειρότερο που θα μπορούσαμε να έχουμε θα ήταν μια έκθεση που δεν θα έχει ευρεία υποστήριξη αλλά για να εξεύρει η υποστήριξη η έκθεση αυτή από ανθρώπους όπως εγώ, ο κ. Φιέλνερ και άλλοι, θέλουμε να είναι φιλόδοξοι. Ο στόχος της παρούσας Επιτροπής είναι η προστασία των καταναλωτών και η αύξηση, η ενίσχυση της νέας αγοράς. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ένα συνολικό πλαίσιο ρύθμισης των επιγραμμικών τυχερών παιχνιδιών που να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά ε, προσώπων που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες με νόμιμο τρόπο. Και να ξεφύγουμε από τους παράνομους operator. Και έτσι να προστατευτούν οι καταναλωτές. Είναι κάπως παράδοξη η θέση μου, με την έννοια ότι επικρίνω ορισμένα μέλη της παρούσας Επιτροπής, διότι μιλούν υπερβολικά για την επικουρικότητα με ιδιαίτερο ζήλο και ενθουσιασμό, διότι πολύ συχνά στην παρούσα Επιτροπή οι συντηρητικοί του Ηνωμένου Βασιλείου ε, βρίσκουν ιδιαίτερα ελκυστική την αρχή της επικουρικότητας για να προστατεύσουν την κυριαρχία της χώρας τους και τότε επικρινόμαστε από τους πράσινους ιδίως, ενώ τώρα ξαφνικά αποφασίζουν οι πράσινοι ότι είναι καλή αρχή της επικουρικότητας γιατί θέλουν να προστατεύσουν τα κρατικά μονοπόλια στις χώρες τους. Ωστόσο, εάν καταστήσετε παρόν, παράνομη την δραστηριότητα αυτή, δεν την εξαφανίζετε, απλώς την κάνετε να περάσει στη μαύρη. Θα πρέπει να είστε σαφείς και σταθεροί απέναντι σε ορισμένα μέλη της παρούσης επιτροπής που θεωρούν ότι όταν κάτι δεν τους αρέσει πρέπει να γίνει παράνομο. Μα δεν σταματά έτσι όμως το επιγραμμικό παιχνίδι είναι παράνομο στη Γερμανία. Ωστόσο, εκτιμώνται σε 2 εκατομμύρια οι Γερμανοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τι υπηρεσίε αυτέ, κάνουν το παιχνίδι αυτό και είναι εντελώ απροστάτευτοι. Έτσι λοιπόν, αν μπορέσετε να καταλήξετε σε κάποιε καλέ συμβαστικέ λύσει που να μπορούν να τι υποστηρίξουν όλοι, τότε θα είμαστε σύμφωνοι. Και σα εύχομαι καλή ε, επιτυχία στι προσπάθειέ σα. Σαφώ το τυχερό παιχνίδι έχει πραγματικά σημαντικές και παράξενες θα έλεγα ας πούμε συνέπειες ε, στη δημιουργία κάποιων ασυνήθιστων ε, συνασπισμών μέσα στο κοινοβούλιο μεταξύ των διαφόρων πολιτικών σχηματισμών. Η κυρία δεν έχω υποβάλει τροπολογίες διότι βρίσκω σωστή την προσέγγιση Κρότσμαν και την υποστηρίζω. Γιατί και εγώ έχω πιστεί ότι πρέπει κάτι να γίνει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ είπα για πολύ καιρό όχι. Είναι θέμα καθαρά των χωρών μελών. Κάτι που λησμονεί ο κύριος Φόξ όπως και άλλοι συναδελφοί μας είναι ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές παραδόσεις σε ό,τι αφορά το παιχνίδι και την αντιμετώπιση του τυχερού παιχνιδιού. Και εγώ θέλω να ληφθεί υπόψη αυτό. Και γι' αυτό τάσομαι εν προκειμένου υπέρ της επικουρικότητας, η οποία όμως δεν αρκεί χρειαζόμαστε και μία ρύθμιση στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Με πείσατε λοιπόν, βρήκα την πρότασή σας άλλωστε λογική και θα σας υποστηρίξω και με τις ε, τροπολογίες ώστε να μην αποδυναμωθεί η ε, πρότασή σας αλλά να παραμείνει ως έχει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Διγιόμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι καλό να λάβουμε υπόψη μας όλες τις πλευρές. Ακούσαμε τη γνώμη της μίας πλευράς, να ακούσουμε και τη γνώμη της άλλης. Σημερίζομαι την ανάλυση σας και θα προσπαθήσω να διευκρινίσω αυτήν την άλλη πλευρά. Το επιχείρημα που λέει ότι δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα, αυτό δεν το συμμερίζομαι. Αν δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να το ευνοήσουμε ε, επιτρέποντάς το εν μέρη. Σε ορισμένες χώρες είναι δυνατόν να στοιχηματίζει κανείς online και δεν διαπιστώνω να μειώνεται η παράνομη προσφορά από την άλλη. Δηλαδή το να νομιμοποιήσουμε εν μέρη δεν επιτρέπει ότι καταπολεμούμε την παρανομία. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη προσφορά. Το συμμερίζομαι αυτό που υπόθηκε για τις πιστοτικές κάρτες. Ναι, μπορούμε να ενθαρρύνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, να έχουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, σύμφωνη. Αν θέλετε να καταπολεμήσετε το πρόβλημα, μπορείτε να συζητήσετε για τις δυνατότητες που υπάρχουν για νόμιμη προσφορά. Πάντως εγώ δεν είδα να... κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα στις χώρες εκείνες οι οποίες επιτρέπουν εν μέρη τον τζόγο διότι εδώ διατρέχουμε τον κίνδυνο να δημιουργήσουμε μία αγορά. Θα κοιτάξω τις τροπολογίες και θα κοιτάξω να σας υποστηρίξω όσο περισσότερο μπορώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αράντ, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε, για την Λυπούμε κύριε Πρόεδρε για την καθυστέρηση. Φυσικά και θα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κρόιτσμαν για το κείμενο αυτό και πρέπει να πω ότι ναι, χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη. Όλοι μίλησαν γι' αυτό και οι, οι σκιώδεις Και το ΕΛΚ θεωρεί ότι η προστιθέμενη αξία της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα είναι πάρα πολύ σημαντική. Καλύτερη προστασία του καταναλωτή, πολέμηση της εγκληματικότητας, διαφύλαξη του αθλήματος. Όπως είπε και η κυρία Σαρμόζερ, ε, αυτή η αγορά δεν είναι μία αγορά όπως οι άλλες. Πρέπει να βρούμε μία ισορροπία, μία ρύθμιση και ένα άνοιγμα. Τέσσερα σημεία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που στο κείμενο και στις πολλές τροπολογίες που κατατέθηκαν η αρχή όχι της παθητικής επικουρικότητας αλλά της επικουρικότητας, της δυναμικής επικουρικότητας υπογραμμίζεται. Το υπογραμμίζει εξάλλου και ο εισηγητής. Όπως το είπαν και προλαλήσαντες υπάρχουν τέτοιες εθνικές διαφορές που αν θα θέλουμε να προχωρήσουμε η ενεργητική επικουρικότητα δεν θα πρέπει να αποτελεί τροχοπέδι, θα πρέπει να αποτελεί μοχλό για να προχωρήσουμε. Αμοιβαία αναγνώριση. Θέλω να επιμένω σε ένα σημείο, το ανέφερα και στην πρώτη ακρόαση, το θέμα της ακαιρεότητας του αθλήματος. Αυτά που λέγονται για την προστασία των καταναλωτών είναι πολύ σωστά, αλλά και η ακαιρεότητα του αθλήματος αποτελεί ένα θέμα Ευρώπης. Πρέπει να προχωρήσουμε στον τομέα, των, στον τομέα αυτών. Είναι ένα στίχημα το οποίο θα πρέπει να θέσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Επιτροπή πιο συγκεκριμένα. Για μας είναι κάτι το θεμελιώδες ε, για την αναζήτηση του συμβιβασμού σε αυτό το κείμενο. Για το θέμα των αδειών είμαι και είμαστε υπέρ της ιδέας της απλούστευσης, διότι η απλούστευση μπορεί να ε, καθιστά και την προσφορά πιο θελκτική. Αποδυναμώνει την παράνομη προσφορά, αλλά τι είναι αυτές οι απλουστευμένες άδειες. Μειώνονται τα διοικητικά βάρη, οπότε συμφωνώ, αλλά ποιος είναι ο τελικός στόχος. Ε, θέλουμε να αυξήσουμε τις άδειες ε, γιατί δεν πρόκειται απλώς εδώ για θέμα αυταρέσκειας. Θα πρέπει φαντάζομαι να υποθεί αν πρόκειται για μείωση του διοικητικού βάρους. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα δεν είναι ίσως η ώρα, αλλά θα θέλαμε να συζητήσουμε για το θέμα. Η θέση του ΕΛΚ για αυτήν την έκθεση, πέρα από τις εθνικές ιδιαιτερότητες που καταγράφονται στις τροπολογίες ορισμένων συναδέλφων, ε, θέλω να σας πω ότι αυτή η θέση είναι μία θέση που συμμερίζονται το μεγαλύτερο μέρος του ΕΛΚ. Εμείς ε, θέλουμε, θα, θα προσπιστούμε δύο βασικούς άξονες, ενεργητική επικουρικότητα, άνοιγμα της αγοράς και ρύθμιση. Να ξέρετε πάντως, για μας, για το ΕΛΚ, εμείς του ΕΛΚ μάλλον θα αναζητήσουμε αυτή την ισορροπία και θα αναζητήσουμε και τον συμβιβασμό γύρω από αυτά τα σημεία. Τελευταίο τώρα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα θετικό μήνυμα προς την Κομισιόν. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι η έκθεση αυτή πρέπει να είναι μια χρήσιμη έκθεση που να αποδεικνύει και στην Κομισιόν ότι τελικά το Κοινοβούλιο δεν είναι ουραγός αλλά είναι, βρίσκεται στην πρωτοπορία, προτείνει, δεν θέλει πισωγυρίσματα, θέλει προχωρήματα προς ευρωπαϊκές θέσεις για να αποδείξει και στον κόσμο ότι τελικά αξίζει τον κόπο. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις και για τα σχόλια τροπολογιών. Ο κύριος Ντεκάμπος και ο Άνδρου Σβάμπ θέλουν το λόγο. Υπάρχει κάποιος άλλος που ζητάει το λόγο. Ο κύριος Ντεκάμπος πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κρόιτσμαν για την εργασία του και να τον συγχαρώ για τον τρόπο με τον οποίο προέβαλε τις προτάσεις του. Κατά απόλυτα σαφή τρόπο και διαφανή και μίλησε για τα πραγματικά ε, διλήμματα τα οποία μας απασχολούν. Υπάρχουν τρία σημεία στα οποία θα ήθελα να σταθώ, την ε, πρόσφατη νομολογία του ΔΕΚ και τα εθνικά μονοπόλια. Ορισμένα κράτη-μέλη μπορούν να κρατήσουν ε, αυτά, αυτή την υποδομή έτσι ώστε να μπορέσουν να καταπολεμήσουν την απάτη και την ε, φοροδιαφυγή. Έχουμε λοιπόν την πάγια νομολογία του ΔΕΚ, αλλά μιλάμε και για περιορισμό των φορέων και ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της μη διάκρισης. Επίσης, μιλάμε για την ανάγκη της διασφάλισης αυτών των υπηρεσιών, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούν να προβληθούν. Τέλος, Όλοι γνωρίζουμε ότι τα online τυχερά παιχνίδια είναι ένας περίπλοκος τομέας και η απελευθέρωσή τους δεν είναι ύψης της σημασίας για την ενία αγορά. Δεν μπορούμε βεβαίως και να στρουθοκαμιλίζουμε και να θεωρήσουμε ότι δεν υφίσταται το θέμα. Βεβαίως η εικονική επικοινωνία άλλαξε τα δεδομένα αυτής της αγοράς και δημιούργησε διάφορους κινδύνους. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ένα ασφαλές πεδίο εφαρμογής διατηρώντας και μάλλον προωθώντας και την ασφάλεια του καταναλωτή πρωτίστως. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλος σε αυτό το γύρο, κύριο Σφάμπ. Ευχαριστώ. Πρώτα θα ευχαριστήσω τον κύριο Αμπάντ για την προσπάθεια που καταβάλει. Τα όσα λέχθηκαν προηγουμένως από τον Ashley Fox είναι απόλυτα σωστά. Τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια είναι σήμερα στην Ευρώπη μια πραγματικότητα η οποία ξεπερνά τα σύνορα των διαφόρων χωρών και δεν έχει νόημα να κλείνουμε τα μάτια μας. Γι' αυτό και εδώ ο Φόξ έχει δίκιο ότι η επικουρικότητα και μόνη της δεν μπορεί να είναι η μόνη πηξίδα που θα ακολουθούν οι χώρες μέλη. Δεν έχει καμιά σχέση αυτό βέβαια με απελευθέρωση. Χρειάζεται περισσότερος έλεγχος μιας αγοράς που όπως είπε και ο εισηγητής κατά επανάληψη είναι αρκετά ανεξέλεγκτη. Το ερώτημα είναι θα αρκεστώ όμω εδώ να κάνω μόνο μια ερώτηση στον εισηγητή, γιατί εγώ δεν είμαι σκιώδη εισηγητή. Εάν όντω εξυπηρετούμε τον στόχο μα, εάν βάλουμε ελάχιστε απαιτήσει, ενώ έχουμε 27 διαφορετικά καθεστώτα με τις ελάχιστες απαιτήσει προκαλούμε τη δημιουργία νέων 27 διαφορετικών καθεστώτων και δεν αλλάζει τίποτα από τη ουσίες. Μήπως είναι καλύτερα να δοθεί στους providers η δυνατότητα να επιλέξουν αν θα ζητήσουν και θα αποκτήσουν εθνική άδεια λειτουργίας ή εναλλακτικά να τους διαθέσουμε, να θέσουμε δηλαδή στη διάθεσή τους ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο όμως θα συνοδεύεται από υψηλές απαιτήσει προστασίας του καταναλωτού και θα λαμβάνει υπόψη βεβαίω ε, και τα συμφέροντα των διαργανωτών των διαφόρων παιχνιδιών και τα σχετικά στοιχήματα από τις χώρες μέλη και εκεί αγαπητέ Fox δεν είμαι βέβαιος αν υπό τις συνθήκες αυτές θα ήσασταν όντως σύμφωνος με ένα τέτοιο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ίσως εκεί ε, να βρίσκεται και η πεμπτουσία της συμφωνίας που μπορούμε να κάνουμε και νομίζω ότι πράγματι η πρόταση Κρότσμαν εδώ είναι η μόνη η οποία δίκησε κάποια λύση. Όπως είπα, ελάχιστες απαιτήσει. Ναι, κύριε Κρότσμαν, μπορείτε να απαντήσετε σε λίγο. Εγώ έχω κάποιες επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά ελάχιστες απαιτήσει από πλευράς χωρών μελών. Πάντως ελπίζω ότι θα μπορέσει να προωθηθεί το θέμα και να ληφθούν αποφάσεις στους επόμενους μήνες. Θα παρακαλέσω την εκπρόσωπο της Κομισιόν να πει λίγα λόγια πρώτα και μετά είμαι σίγουρος ότι ο κ. Κρόισμαν θα θέλει να δευτερολογήσει. Θα έχουμε κάποιο χρόνο ακόμη ώστε να μπορέσουν να παρέμβουν και άλλοι εάν προκύψουν θέματα από την παρέμβαση της Κομισιόν. Και απρόμπτω. και ίσως να μας δώσει και κάποιες ε, πληροφορίες σχετικά με το ποιες είναι οι σκέψεις επί του παρόντος της Κομισιόν για το θέμα αυτό. Διότι ακόμα στην Πράσινη Βίβλο δεν έχει ε, ταχθεί υπέρ καμιάς λύσεω. Μήπως θέλει να μας αποκαλύψει κάποια από τα μυστικά των σκέψεων της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόιτσμαν για την πληρότητα και τη φιλοδοξία της έκθεσης του βλέπουμε ότι όλα τα θέματα που θίξαμε στην πράσινη βίβλο ε, φύγονται και στην έκθεση και προτείνονται και λύσεις για το μέλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες που δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέλη της Επιτροπής και ότι υπάρχει μία σύγκληση σε σχέση με την προσθέμενη αξία της δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός είναι ο βασικός ε, μας στόχος, δηλαδή να καταπολεμήσουμε τις παράνομες προσφορές και να προωθήσουμε μία πολύ καλή πλαισίωση, ποιοτική πλαισίωση για, την επιγραμμική, για τα επιγραμμικά τυχερά παιχνίδια. Βεβαίως υπάρχουν πολλά επιμέρους ζητήματα όπου υπάρχουν αποκλήσεις. Μιλάμε για συνεργασία μεταξύ κρατών μελών που μπορεί να οδηγήσει σε μία πλήρη οδηγία που να καλύπτει το όλο ζήτημα. Για την Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική η τελική έκβαση της έκθεσης, διότι θα μας ορίσει την κατεύθυνση που θα πρέπει να λάβουμε μετά από την Πράσινη Βίβλο. Ε, ρωτήσατε κατά πόσο υπάρχουν δεδομένα, θα σας απογοητεύσω γιατί βρισκόμαστε σε φάση διαβούλευσης, δεν φτάσαμε σε συμπεράσματα. Βρισκόμαστε στο πέρας της διαδικασίας διαβούλευσης. Έχουμε λάβει 250 απαντήσεις που δεν φαίνονται πολλές εκ πρώτης όψεως, αλλά πρόκειται για μεγάλους φορείς, για σημαντικούς φορείς, Και υπάρχουν και οι μεσάζοντες που είναι πολύ σημαντικοί. Μιλάμε για πάροχους διαδικτύου και πάροχους υπηρεσιών. Απάντησαν όλοι Μιλάμε και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων, την καταπολέμηση της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και γι' αυτό θα πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε αυτές τις 250 απαντήσεις και να μπορέσουμε να συντάξουμε μία έκθεση που θα δώσει μία μακροχρόνια πορεία, η κατεύθυνση προς το μέλλον. Άρα σήμερα δεν είμαι σε θέση να σας δώσω στοιχεία. Σίγουρα στην Ολομέλεια η Επιτροπή θα είναι σε θέση να πει πολύ περισσότερα. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κυρία Μπρόντε δεν αποθαρρυνόμαστε από την απάντησή σας, διότι πιέζεται ακόμα περισσότερο τον κύριο Κρόιτσμαν να φτάσει σε δόκιμες λύσεις. Εάν το Κοινοβούλιο φτάσει σε μία συνένεση, τότε η Επιτροπή θα έχει άλλη θεώρηση, θετική θεώρηση. Βεβαίως, ε, μέσα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας σας μπορείτε να κινηθείτε όπως θέλετε. Κύριε Κρόιτσμαν, τι έχει να μας πείτε σε σχέση με τα όσα ακούσατε μέχρι τώρα και αν υπάρχει και κάποιος άλλος που θα ήθελε να λάβει το λόγο μπορεί να το κάνει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο στόχος μου είναι να επιτύχω ευρία πλειοψηφία υπέρ των αδειών. Επειδή η κυρία Σαλεμόζε δεν θα συμφωνήσει, δεν θα μείνουμε στην επικουρικότητα. Και η Κομισιόν θα κινηθεί, θα παραμείνει σε αυτά που έχει μέχρι τώρα, διότι διότι κάθε χώρα μέλος θα προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει τα έσοδά της χωρίς να προβεί στην χορήγηση αδειών. Ενώ για μένα η χορήγηση αδειών είναι στην πραγματικότητα έκφραση μιας ενεργού επικορικότητας. Την επικορικότητα δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Μπορούμε να πούμε ότι θα φτιάξουμε ένα πλαίσιο και αυτό θα είναι όλο. Δηλαδή την τελευταία απόφαση την έχουν όντως οι χώρες μέλη. Άρα έρχομαι τώρα στον κύριο Σβάπ. Οι απαιτήσει τι οποίε αναφέρθηκα δεν θα είναι ελάχιστε απαιτήσει. Είπα ότι θα φτιάξουμε ευρωπαϊκές απαιτήσει καταπολέμηση των απατών, καταπολέμηση του εθισμού στο παιχνίδι κλπ. Και οι χώρες μέλη μπορούν να επιβάλλουν παραπάνω και τότε θα αποφασίσουν οι χώρες, κυρία Σαλδεμόζη, αν θα διατηρήσουν τα μονοπόλια ή όχι. Εγώ γνωρίζω την νομοθεσία του Σλέσι Χολστάιν που λέει το λότο εξακολουθεί και είναι κρατικό. Όλα τα άλλα μπορούν να υπαχθούν σε κάποια κανονιστική ρύθμιση. Το λότο μπορεί να γίνει τότε και επιγραμματικά, και επιγραμμικά μάλλον. Ε, το ίδιο για τα καζίνο. Άρα χρειάζεται έκδοση και χορήγηση ε, αδειών. Χρειαζόμαστε όμως ευρεία πλειοψηφία, διότι κυρία Σάλντε Μόζε, εάν δεν τα ζητήσουμε όλοι μαζί, τότε θα δούμε την Ευρωπαϊκή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην κινείται. Και η κυρία της Κομισιόν μόλις τώρα μας εξήγησε, μας δήλωσε προς τα που θα πάει. Αν δηλαδή το Κοινοβούλιο δεν συμφωνήσει, δεν, ε, είναι, ο, ε, δεν είναι ενωμένο, τότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ας το λάβουμε υπόψη αυτό, να δούμε δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να σπρώξουμε την Κομισιόν για να κάνει κάτι. Μόνο εφόσον εδώ εξασφαλίσουμε ευρεία πλειοψηφία και να δούμε τότε αν θα μπορούμε να είναι κάπως πιο φιλόδοξη η νομοθετική αυτή ρύθμιση ή όχι. Ελάχιστες ε, απαιτήσει κύριε Σφάπ δεν σημαίνει πραγματικά ελάχιστες και μετά όπως είπε ο κύριος Σαμπάτ μπορούμε να κάνουμε τη ρύθμιση. Εάν μια χώρα μέλος πει ότι μου αρκεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο, προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή για να προβώ στην ε, χορήγηση αδειών, έχει καλώς. Είμαστε σύμφωνοι. Εάν όμως θέλει να αυξήσει τι απαιτήσει επίση είναι εντάξει. Επίση υπάρχουν ορισμένε τροπολογίε οι οποίε αφαιρούν τη λέξη ελάχιστε από τι απαιτήσει και παραμένουν μόνο οι απαιτήσει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά βέβαια δεν θα το επιτρέψει η επικουρικότητα. Δεν έχει νόημα να παίρνουμε φόρα και να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο οι Μαλτέζοι ήρθαν και μου είπαν, αν λοιπόν έχουμε έγκριση λειτουργίας στη Μάλτα, τότε θα μπορούμε να έχουμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι. Όχι, έτσι δεν θα λειτουργήσει. Θα πρέπει να έχουν ωστόσο όλη τη δυνατότητα να να, να ε, πληρούνται και οι προθυποθέσεις της ε, νομοθεσίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και όχι όπως ε, οι Γερμανοί που νομίζουν από τους εκατοντάδες που θα υποβάλουν αιτήσει για χορήγηση αδειών θα μπορέσουν να επιλέξουν μονάχα 6-7. Το ίδιο συμβαίνει στο κρατήριο του Σλέσβι Χόλσταϊν. Δεν μιλούμε για αυτό όμως, δεν μιλούμε δηλαδή για κρατικές ρυθμίσεις. Θα παρακαλέσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους που θέλουν αυτή την ενεργοεπικουρικότητα να ταχθούν υπέρ της οδηγίας και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει οδηγία. Και τότε όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι γιατί θα έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Μια στιγμή, αν μου επιτρέπετε να απαντήσω πρώτα και μετά να έρθουμε στο χρονοδιάγραμμα. Α, κυρία Σαλντεμόζε. Θα προσπαθήσω να τα πω στα αγγλικά αυτή τη φορά, ώστε να είμαι βεβαίω ότι θα με καταλάβετε καλά. Και θα σας το πω καθαρά. Δεν υπεραμείνομαι των κρατικών μονοπωλίων, ούτε εγώ ούτε η πολιτική μου ομάδα. Υποστηρίζουμε το δικαίωμα των χωρών μελών να καθορίζουν τις αγορές τους τυχερών παιχνιδιών. Αν η Γερμανία θέλει μονοπόλιο, έχει καλά. Το δανεικό μοντέλο είναι license model, με άδειες δηλαδή. Αλλά και το βρίσκω καλό. Δεν θα ζητήσω όμω από όλε τι χώρε τη Ευρώπη να υιοθετήσουν το δανεικό μοντέλο. Αυτό που θέλω να πω με λίγα λόγια είναι ότι δεν έχω αντίρρηση για αυτή την ενεργό επικουρικότητα που λέτε. Από την άλλη μεριά όμω πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ακολουθούμε τον ίδιο ορισμό. Η επικουρικότητα είναι σημαντική για μένα. Ναι, μεν ενεργό, να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι τι στο ευρωπαϊκό επίπεδο, και εγώ συμφωνώ μαζί σα. Αλλά τι είδου δράση θα αναλάβουμε, αυτό είναι το ερώτημα. Ο κύριο Σαμπάτ είπε ότι δεν είναι βέβαιο ότι έχει έρθει ο χρόνο για να υπάρξει πραγματικά οδηγία. Και εγώ συμφωνώ μαζί του. Αυτό πρέπει να κάνουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ασφαλώ και είναι κάτι που πρέπει να στηρίξει, να ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών. Το ερώτημα όμω είναι πώ. Ακριβώς, όχι αυτό που λέτε. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αρχίσουμε να αναζητήσουμε ένα τρόπο καλύτερη συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών. Να φτιάξουμε ένα είδος πλαίσιο δηλαδή. Δεν ζητώ ευθύ αμέσω οδηγία. Μπορεί να χρειαστούν 2, 3, 5, 10 χρόνια. Δεν είμαι αντίθετη, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι όριμος ο χρόνος σε κάτι τέτοιο τώρα. Μη λέτε όμως, μη με κατηγορείτε όμως ότι δίθεν δεν θέλω να γίνει τίποτα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι αυτή η θέση μου. Εγώ θέλω κάτι να κάνουμε. Αλλά θέλω να γίνει το σωστό για την ώρα. Και δεν νομίζω το σωστό είναι τώρα οδηγία. Και για να είμαστε ειλικρινεί, γνωρίζουμε όλοι ότι η μεγάλη δυσκολία θα αντιμετωπιστεί στο Συμβούλιο, γιατί οι περισσότερες χώρες μέλη δεν θέλουν να υπάρξει ευθύ αμέσω οδηγία. Α προχωρήσουμε λοιπόν βήμα-βήμα και ίσω σε κάποια χρόνια ε, να βγω κι εγώ να, και να υποστηρίζω την ιδέα μια οδηγία. Ωστόσο, μην με κατηγορείτε ότι δεν θέλω ε, ευρωπαϊκή λύση ή δεν θέλω να γίνει. Όχι, γιατί κάπω θύμωσα με αυτά που είπατε. Εγώ δεν στηρίζω τα κρατικά μονοπόλια. Ούτε υποστηρίζω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε τίποτα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήθελα λοιπόν να σα το ξεκαθαρίσω απολύτω αυτό. Αν καταλάβετε την βάση των λεγόμενων μου τώρα, τότε νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση. Μια φράση μόνο, κύριε Πρόεδρε. Το πρόβλημα είναι το εξή, λέει ο κύριος Κρόισμαν. Εάν δεν κάνετε τίποτε, εάν δεν συνεργαστούμε, δεν θα γίνει τίποτε. Και βεβαίω το δεύτερο που λέτε έχετε δίκιο. Εάν ε, κάνετε οδηγία στο ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται τη συνεργασία του Συμβουλίου. Είδατε όμω ότι υπάρχουν και μεγάλε διαφορέ και ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα συμβασμό. Γι' αυτό λέω να φτιαχτεί ένα πλαίσιο όπου οι διάφορε χώρε μέλη να μπορούν να προσθέσουν κάτι. Και αυτή θα είναι η καλύτερη λύση. Να γίνει κάτι που να μπορούν να το δεχτούν όλοι, γιατί αλλιώ δεν πρόκειται να υπάρξει πλειοψηφία στο Συμβούλιο. Για μένα είναι σαφέ ότι η έκβαση προς την πλευρά της οδηγίας δηλαδή είναι ανοιχτή διότι χρειάζεται η συνεργασία του Συμβουλίου. Και γι' αυτό είπα ότι για μένα ασφαλώς είναι, είναι απαραίτητο για μας το Συμβούλιο. Θα δούμε τότε όμως ποια θα είναι η έκβαση της οδηγίας. Να υπάρχει όμως το, το, το πλαίσιο όπου να μπορούν αναλόγως με διαφορετικές παραδόσεις κτλ. οι χώρες να προσθέτουν απαιτήσει. Νομίζω ότι χρειάζεται κάπως περισσότερη συνεργασία και βεβαίω, αν γίνει αυτό και υπάρξει η πλειοψηφία, θα πρέπει να γίνει δεκτή και από το Συμβούλιο. Ωραία είναι ε, να μιλούμε αγγλικά και να κάνουμε συζητήσεις που θα είναι πιο παθιασμένες τότε. Ο κύριος Μάιερ που δεν έχει μιλήσει προηγουμένως. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ έχω υποβάλει ορισμένε τροπολογίε. Ο εισηγητή και δικαίω από την πλευρά του είπε ότι δεν συμφωνώ με την άποψή του. Για διάφορους λόγους. Μετά τα όσα λέχθηκαν τώρα θα πρέπει να σκεφτώ ξανά την θέση μου αν είναι λογική. Αλλά έχουμε 27 χώρες μέλη με 27 διαφορετικές παραδόσεις για το τι είναι τυχερό παιχνίδι. Αυτά δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να εννοποιηθούν. Δεύτερο, εάν επιβάλλουν μια οδηγία με απαιτήσει, για παράδειγμα, για την χορήγηση αδειών, θα δείτε ότι θα ξεκινά μια κίνηση που θα αναγκάσει κάθε χώρα να χορηγήσει άδειε, ακόμη και αν δεν θέλει. Θα υπάρξει τότε αυτομάτως μια ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο απέτηση για τη χορήγηση αδειών. Μην το λησμονείτε αυτό. Μια οδηγία περιλαμβάνει και μια υποχρέωση, αλλά αποτελεί και τη βάση για απαιτήσει. Εκεί λοιπόν έχω τις μεγάλες μου ε, επιφυλάξεις. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά πράγματα που ήθελα να πω για την ώρα. Το τελικό θέμα όμως σχετίζεται με, το, με αυτό που είπε και ο κύριος Φόξ. Οι εξελίξεις των επιγραμμικών τυχερών παιχνιδιών σε σχέση με τη συμμετοχή των καταναλωτών άλλαξε το τοπίο των παιχνιδιών αυτών στο Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το σημείο εκκίνηση. Τώρα, τι κάνουμε. Η κυρία Σάλτε Μόζε είναι πολύ ρεαλίστρια διότι τόνισε το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να προβάλλουν μια συνολική λύση. Όμως έχουμε να κάνουμε και με θέμα προστασίας των καταναλωτών, γιατί πολλές φορές απαγορεύουμε τη, τα επιγραμμικά στοιχήματα, αλλά στην ουσία είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα πρέπει να προβάλλουμε μια συνετή λύση. Θα πρέπει να δεχτούμε το γεγονός ότι η κατάσταση αλλάζει. Και αυτό είναι ε, δύσκολο βεβαίως, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε πραγματιστές. Και νομίζω ότι και οι πολίτες θεωρούν ότι πολλές φορές ε, δεν είμαστε ρεαλιστές όταν απαγορεύουμε. Και αυτό στην ουσία υποσκάπτει οποιοδήποτε δικαιοδοτικό σύστημα, διότι οι καταναλωτές πολίτες έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αλλά σε ορισμένες χώρες είναι παράνομο να έχουν κέρδη. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν στην πλευρά του πολίτη, όπως και να έχει. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Νομίζω ότι έχετε τις ε, πληροφορίες. Μπορείτε να το αναφέρετε εσείς. Από όσο βλέπω θα ψηφίσουμε στις 19 Σεπτεμβρίου Νομίζω ότι θα γίνει και μία συνάντηση. Είμαστε... Ε, δεν ε, διαφέρουμε τόσο πολύ με την κυρία Σάλντε Μόζε. Και θα πρέπει να αποφασιστεί τι θα γίνει για να υπάρχει μια πλειοψηφία. Είναι δική μας αυτή η έκθεση, άρα δεν έχουμε χρονική πίεση. Αν χρειαζόσαστε περισσότερο χρόνο για ένα καλύτερο αποτέλεσμα, τότε εμείς δεν θα αντιταχθούμε. Ίσως βεβαίως θεωρήσετε ότι θα πρέπει να αρκεστείτε στις 19 ε, Σεπτεμβρίου. Αυτό μπορείτε να το ε, αφήσετε στην Ολομέλεια, δηλαδή να φτάσουμε σε συμβιβασμούς μετά την Επιτροπή. Όπως είπε και η κυρία Ρουλέ, σε διαφορετική περίπτωση θα το συζητήσει στην ομάδα της. Για μένα δεν είναι πρόβλημα. Ας προσπαθήσουμε να αρκεστούμε στο χρονοδιάγραμμα και αν σταθεί αναγκαίο θα παρατείνουμε. Δεν θα ήθελα μετά την ψηφοφορία της Επιτροπής να έχουμε πολλές τροπολογίες στην Ολομέλη, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν εργαστήκαμε καλά και αυτό με απογοητεύει ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και πολλές φορές η διάσκεψη των Προέδρων αναπέμπει το θέμα στην Επιτροπή. Εσείς είσαστε εμπειρογνώμονες είσαστε ο εμπειρογνώμων, γι' αυτό θα πρέπει να το επιλύσουμε εμείς. Δείτε το στις πολιτικές ομάδες για να μην φανεί ότι δεν εργαστήκαμε παρκώς. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε καλή ποιότητα για να φτάσουμε σε καλά αποτελέσματα. Δείτε το με τους σκιώδεις και αν έχετε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα θα το δούμε στη διάσκεψη των Προέδρων έτσι ώστε να βρούμε ένα άλλο σλότ ε, στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι η κυρία Μπρόμπτε θα πρέπει να ε, μας απαντήσει και όλα στην Ολομέλεια, δηλαδή η Επιτροπή όχι ίδια. περισσότερες ε, τροπολογίες θέλουν να δώσουν ουσιαστικό χαρακτήρα στην έκθεση. Θα πρέπει να αποφασίσουμε κατά πόσο θα ε, θέλαμε να έχουμε μία οδηγία ή όχι. Υπάρχουν και θέματα ίσονος σημασίας, αλλά δεν αποτελούν πρόβλημα. Αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί. Εγώ θα προτιμούσα να έχουμε μεγάλη πλειοψηφία, αλλά και μικρή να έχουμε καλός. Γιατί στη δική μου ομάδα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις αναχώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως είπε και η κυρία Σάλντε Μόζε και ο κύριος Αράντε, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ίσως το επιλύσουμε σε επίπεδο, σε σκιωδών. Okay, well, Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες. Ας ελπίσουμε να έχουμε πολλές παρόμοιες. Έχουμε και την τελευταία μας έκθεση σήμερα δηλαδή ένα σχέδιο γνωμοδότης του κυρίου Φερνάντο Ντεκάμπος. Μία δική μας γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων σε σχέση με συγκεκριμένες κρατικές ενισχύσεις σε σχέση με, που να ισχύουν για τις ΔΕΚΟ. Ο κύριος Σβάμπ είναι σκιώδης από το ΕΛΚ. Ο κύριος Κρόιτσμεν για τους φιλελευθέρους. Από τους πράσινους ποιος είναι παρόν. Ο κύριος Διόν θέλει να είναι σκιώδης. Εγώ είμαι από, την, από τους Ευρωπαίους ε, συντηρητικούς. Καλωσορίζω και την Επιτροπή κυρία Γκικόπεν θα μας απαντήσει σε σχέση με, τα, με όλα τα θέματα, με όλα τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν αυτή τη μεταρρύθμιση. Ο κύριος Κορέια Ντεκάμπος έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ καταρχήν θα πρέπει να πλαισιώσουμε τις ΔΕΚΟ, να θυμίσουμε την ιστορική τους πορεία. Αυτές οι υπηρεσίες προέκυψαν σε μία φάση όπου δεν υπήρχαν ε, μέσα της αγοράς και το κράτος έπρεπε να παράσχει όλες τις υπηρεσίες, τις συλλογικέ υπηρεσίες. Γι' αυτό προέκυψαν οι δέκο για οικονομικούς ή κοινωνικούς σκοπούς για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Δυστυχώς υπήρξαν πολλές ελλείψεις της αγοράς και γι' αυτό το κράτος έπρεπε να επέμβει. Θα έπρεπε λοιπόν να καλύψουμε την προσφορά και τη ζήτηση καθώς και τις, ε, τα διάφορα αγαθά και τις υπηρεσίες. Αυτά τα χάσματα της αγοράς έπρεπε να πληρωθούν από την κρατική παρέμβαση με βάση τις καθολικές αξίες, ευρωπαϊκές αξίες. Έτσι ανέκυψαν οι ΔΕΚΟ. Το κείμενο της Κομισιόν καταδεικνύει ότι παρά το γεγονός ότι οι κρατικές ενισχύσεις λειτουργήσαν καλώς, παρόλα αυτά υπάρχουν αμφισημίες ως προς τις κοινωνικές υπηρεσίες και γι' αυτό χρειάζονται νομικές ε, διασαφήσεις και σαφή και αναλογικά μέσα, έτσι ώστε να υπάρχει μια μεγάλη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα καθώς και ποιοτική συνεισφορά των ΔΕΚΟ. Θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογική προσέγγιση όλων των υπηρεσιών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν στρεβλώσεις ανταγωνισμού, ιδιαίτερα ως προς τις ε, διασυνοριακές συναλλαγές. Γι' αυτό προβάλαμε συστάσεις προς την Επιτροπή Οικονομικών υποθέσεων και θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να αναλυφθεί μια νομοθετική πρωτοβουλία έτσι ώστε ε, δυνάμει του άρθρου 14 της συνθήκης και του πρωτοκόλου 26 να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα άρθρα περί ανταγωνισμού 106 και 107 της συνθήκης. Τα κριτήρια επικαιροποίησης των ΔΕΚΟ θα πρέπει να σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της αγοράς και την υπεράσπιση των κοινωνικών προαπαιτήσεων λαμβάνοντας υπόψη την σωστή οριοθέτηση αυτών των υπηρεσιών που να τις διαφοροποιεί από τις δέκο μη οικονομικού χαρακτήρα. Με βάση δηλαδή μία νομική βάση έτσι ώστε να μην γίνονται παραβάσεις ή παραβιάσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, ιδιαιτερότητες ε, λοιπόν σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο με βάση μια διαδικασία απλούστευσης που να προωθήσει τις ΜΜΕ. Περιμένω τις υποδείξεις των συναδέλφων λοιπόν σήμερα ή τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, στις 19 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για όλες τις υποδείξεις καθώς και για τις μελλοντικές προτάσεις τροπολογιών. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φάμπ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως και εισηγητής τώρα πράγματι της ομάδας μου θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και είμαι βέβαιος ότι θα διεξαχθούν ακόμη συζητήσεις για τις λεγόμενες καθολικές υπηρεσίες. Πρώτα, επιθυμώ να πω ότι η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει ορισμένε θετικές πτυχές. για τουλάχιστον τις κοινέ απαιτήσει για μια ελάχιστη ρύθμιση στο τοπικό επίπεδο, την εξέταση το, για τις τιμές κατοφλίου μάλλον για τις αποφάσεις για τις καθολικές υπηρεσίες και ούτω καθεξής. Και νομίζω εν προκειμένου ότι με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενιαία αγορά αλλά και για τις υπηρεσίες καθολικού ενδιαφέροντος μπορούμε να καταλήξουμε σε μια λύση. Σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση του κυρίου Κορέα Τεκάμπος, εδώ θέλω να περιοριστώ σε τρία θέματα όπου θα υποβάλω και σχετικές τροπολογίες. Κύριε Τεκάμπος, εσείς ζητείτε νομοθετική πρωτοβουλία του άρθρου 14 και των άρθρων 106-107 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για λόγους ε, όχι δογματικούς δεν δέχεται η πολιτική μου ομάδα την ε, νομική βάση της παραγράφου του άρθρου 14 και αυτό το δήλωσε και ο Επίτροπος Σαλμούνια μπορεί να γίνει μια διαφορετική ρύθμιση ανακλάδο αλλά βέβαια υπάρχει και η αρχή της επικουρικότητας που μόλις πριν λίγο την επενούσαμε τόσο πολύ και η οποία επιβάλλει ώστε οι χώρες μέλη, στις χώρες μέλη μάλλον, οι αρχές τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης να αποφασίζουν οι ίδιες. Επίσης λέτε στην γνωμοδότησή σας ότι ένας μονοσήματος σαφής ορισμός των υπηρεσιών καθολικού συμφέροντος αλλά και μη οικονομικού χαρακτήρα θα είναι απαραίτητος και σημαντικός. Όντως αυτός ο ορισμός είναι σημαντικός αλλά εξακολουθεί και παραμένει μέσα στη διακριτική ευχαίρεια των χωρών μελών. Μιλήσαμε σήμερα το πρωί για την εναρμόνιση. Για παράδειγμα η ΜΕΑ στο Βέλγιο είναι υπηρεσία καθολικού συμφέροντος στην Γερμανία είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Έρχομαι και στην παράγραφό σας 6 που αναφέρεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα των δημοσίων προμηθειών. Πάλι εδώ πρέπει να δούμε πού βρίσκεται το σημείο τομής μεταξύ των δημοσίων προμηθειών και της εξασφάλισης των υπηρεσιών καθολικού συμφέροντος. Και σε αυτό προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή ελάχιστες προϋποθέσεις μιας ε, de minimis ρύθμισης. Πάντως νομίζω ότι με την κατάλληλη συζήτηση μπορούμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Είναι και το θέμα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου από το 2003 στην περίπτωση Altmark Transval. Και βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι παροχή υπηρεσίας έχει καθολικό χαρακτήρα όταν υπακούει σε τέσσερις προϋποθέσεις. Η εξέταση, εάν ισχύουν αυτές οι προϋποθέσεις, δεν επαφίεται όμως στις χώρες μέλη, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να εξετάσει εάν ε, πληρούνται τα τέσσερα αυτά κριτήρια, τις αυτές προϋποθέσεις για τη χορήγηση κρατικής ενισχύσεως σε μια υπηρεσία καθολικού χαρακτήρα. θα συζητήσουμε με τον κύριο Ντεκάμπος και το θέμα της νομικής βάσης του άρθρου 14 και ελπίζω θα καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριο Σφάπ. Ο κύριο Κρότσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα συγχαίρω και εγώ τον κύριο Ντεκάμπος. Έχει δίκιο που δέχεται την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικό οι υπηρεσίες καθολικού οικονομικού ε, συμφέροντος να υπάρχουν σε ξεκάθαρους κανόνες. Αυτό πρέπει να είναι το αίτημα όλων των ενδιαφερομένων ώστε να καθίστανται προσιτές αυτές οι υπηρεσίες. παρόλες οι ειδικές ρυθμίσεις εξακολουθούν να υπάρχουν θεμελιώδη ερωτήματα που αποτελούν και τα μεγαλύτερα προβλήματα για το μέλλον. Έτσι είναι σαφές στο τοπικό και περιφερικό επίπεδο εάν ε, τι χαρακτήρα δηλαδή είναι τα, ε, οι κρατικές ενισχύσεις που δίνουν τις υπηρεσίες γενικού και οικονομικού συμφέροντος. Πρέπει να γίνει καλύτερη η ενημέρωση για τους υφιστάμενους κανόνες, καθώς επίσης και η δημιουργία του απαραίτητου νομικού πλαισίου. Η διαφοροποιημένη προσέγγιση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου φαίνεται σωστό βήμα. Ωστόσο δεν πρέπει να λησμονείται ο στόχος, δηλαδή καλύτερος ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων της οικονομίας και η σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και για τις ενισχύσει για τις υπηρεσίε γενικού οικονομικού συμφέροντος. Ωστόσο, πρέπει και οι σχετικές δαπάνε και θυσίε των ενδιαφερομένων να είναι ανάλογες. Τέτοιε υπηρεσίε δεν έχουν μεγάλη συνέπεια στο εμπόριο μεταξύ των ε, ε, χωρών μελών. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα ανάμεσα στις προσπάθειες που καταβάλουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές και στο αποτέλεσμα. Χαίρομαι για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μην, που θα εξυπηρετήσουν το, τον ορθό ανταγωνισμό και με ενισχυμένο έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων που δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα συνήθη περιθώρια κέρδους και για άλλους φορείς της οικονομίας την προσφορά υπηρεσιών πρέπει να ισχύουν παρόμοιοι κανόνες. Όποιος εργάζεται αποτελεσματικά πρέπει να ε, επιβραβεύεται. Για τις ε, υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος πρέπει να υπάρχει και κίνητρο ώστε να διασφαλίζεται και η καλή δαπάνηση του δημοσίου χρήματος. Αυτά τα έχω ε, υποβάλει και ως τροπολογίες που ελπίζω να ληφθούν υπόψη. Θα υποβάλω μάλλον τροπολογίες. Και ευχαριστώ και πάλι για την εργασία του κ. Δεκάμπος. Κανένα από τους πράσινους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη γνωμοδότηση αυτή γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος υποβολής ε, τροπολογιών. Όπως είπε και η Κομισιόν, χρειαζόμαστε ορισμένες ε, διασαφήσεις. Υπάρχουν ορισμένες ε, επιφυλάξεις σε σχέση με πρωτοβουλίες νομοθετικού περιεχομένου. Ως προς την απλούστευση, η Επιτροπή ήδη μας υπέβαλε συγκεκριμένες ε, προτάσεις και ιδέες για μία ντεμίνιμης ε, προσέγγιση η οποία είναι πολύ καλή. Η μόνη μου, το μόνο μου ερώτημα ως προς την ανακοίνωση της Επιτροπής είναι ότι κατά το τέλος η Επιτροπή ε, θέλει να ελέγξουμε την ε, αποδοτικότητα σε επίπεδο κρατών μελών ως προς τους κανόνες ανταγωνισμού. Αλλά ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει βεβαίως αιτιώδη συνάφεια με θέματα οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά δεν νομίζω ότι θα ταχθούμε υπέρ. Και νομίζω ότι ο εισηγητής της καθιστά σαφές ότι θα πρέπει να βασιστούμε στους ε, κανόνες ανταγωνισμού και όχι σε άλλους ε, κανόνες. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και να υποστηρίξω τον εισηγητή. Και εγώ εντάχει θα ήθελα να πω ως κοιόδης για την ομάδα μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντώνιο γιατί άνοιξε τη συζήτηση επί του θέματος, αν και υπάρχουν τομείς ε, όπου δεν εστιάζουμε την προσοχή μας αποκλειστικά στην πρόταση της Επιτροπής, αλλά σε άλλα θέματα σε σχέση με τις υπηρεσίες ε, γενικού ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή κατέστησε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες είτε πρόκειται για μονοπόλιο είτε για έναν εμπορικό φορέα είναι θέματα που αφορούν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερους ο... δεν, θα πρέπει, δεν χρειάζεται να έχουμε καλύτερους ορισμούς, διότι τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, Στη χώρα μου οι υπηρεσίες ύδατος αφορούν τον ιδιωτικό τομέα, αλλά με έναν εθνικό ρυθμιστή, ο οποίος ορίζει τα περιθώρια επενδύσεων, κίνησης και ούτω καθεξής. Σε άλλες χώρες υπάρχει είτε κρατικό μονοπόλιο ε, μία καθαρά περιφερειακή προσέγγιση. Άρα ερμηνεύω διαφορετικά το θέμα από τον κύριο Ντιγιόν. Ως προς την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα. Και αυτό από όσο γνωρίζω σχετίζεται με τον ε, ιδιωτικό τομέα με βάση τις κατευθυντήριες ε, γραμμές μέσα στα πλαίσια μιας εθνικής ρυθμιστικής αρχής. Γι' αυτό χρειάζεται δημόσια υποστήριξη έτσι ώστε να μπορεί να δράσει κανείς αποτελεσματικά, αλλά αυτό δεν κινείται με κριτήρια κέρδους καθαρά. Νομίζω ότι η προσέγγιση της Επιτροπής είναι ότι υπάρχει μία αίρα, μία εθνική ρυθμιστική αρχή, υπάρχει έγκριση, αλλά σε έναν ολοένα και εξελισσόμενο κόσμο θα πρέπει να προβάλλουμε νέες λύσεις με βάση οικονομικά κριτήρια και από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μιλάμε μόνο για κρατικά μονοπόλια πλέον. Επίσης ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και ίσως η Χάιντι και άλλοι θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα, είναι να δούμε πώς, έχει, πώς έχουν οι αγορές δημόσιων προμηθειών. Ε, υπάρχουν δηλαδή τοπικές αρχές που θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες και για λόγους ανταγωνισμού πολλές φορές δεν υπάρχει σαφής αντικατοπτρισμός με τους βασικούς κανόνες της αγοράς ε, αγορών στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Άρα αυτό μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι, τι θέλει να κάνει η Επιτροπή και να μην μιλάμε για νέους ορισμούς. Να μην μιλήσουμε δηλαδή για υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Δεν έχει νόημα να το προβάλλουμε αυτό σε αυτή τη γνωμοδότηση. Έχουμε τρεις ομιλητές και μετά θα ήθελα να μιλήσει η Επιτροπή. Κορότσα Μπίλτ, Βάιλερ και κυρία Γιού. Πρέπει να τελειώσουμε στις 6.30. Κυρία Βανιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον Αντώνιο για την ε, συνθετική γνωμοδότηση που συνέταξε. Δεν είναι τόσο εύκολο να καταφέρει κανείς για ένα θέμα σύνθετο σαν και αυτό να πετύχει αυτό που πέτυχε, Αντώνιο. Συμμερίζομαι απόλυτα αυτό το οποίο έγραψε ο Αντώνιος στην παράγραφο 2 και κύριε Σβάπ, μπορούμε να το συζητήσουμε. Όλοι συμφωνούμε για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και το πλαίσιο πρέπει όμως να φανταστούμε ένα κοινό πλαίσιο ποιότητας όπου θορίζουμε τα κριτήρια, του στόχους και τις αξίες που θέλουμε να εμπεριέχουν αυτές οι υπηρεσίες για την εσωτερική αγορά και να διασφαλίσουμε και μία νομική ασφάλεια μέσα από την νομοθετική πρωτοβουλία. Και αυτή είναι δηλαδή και όλη η δυσκολία του θέματος θα αφήνει δηλαδή το πάνω χέρι στα κράτη, μέλη την αρχή της επικουρικότητας θα την κρατήσουμε. Αλλά και πιστεύω ότι θα είναι εφικτό κάτι τέτοιο και βασίζομαι στην Κομισιόν διότι αυτό το οποίο μας προτείνει ο Αντώνιος στη γνωμοδότησή του και μας προτείνει και η Κομισιόν μας δείχνουν ότι μπορούμε να βρούμε μια κοινή πορεία όλοι μαζί. Για την παράγραφο 3 Αντώνιο ε, θα κάνω μία μικροτροπολογία. σύμφωνο με αυτό το οποίο γράφεις. θεωρώ για την αποτελεσματικό ότι, πρέπει να είναι αποτελεσματικές οι αγορές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε τα κοινωνικά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές είναι εμπλεκόμενα μέρη στην αποτελεσματικότητα και στην ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής αγοράς. Η ευημερία των εργαζομένων αλλά και τα κίνητρα που έχουν οδηγούν στο να εκτιμούν την εσωτερική αγορά και να θέλουν να την καταστήσουν ανταγωνιστική. Θέλω να τονιστεί αυτή η πλευρά. Τώρα για τους ορισμούς έχουμε πάντοτε το ίδιο, τον ίδιο διάλογο που δεν καταλήγει ποτέ, αλλά πρέπει να τον συνεχίσουμε. Αυτός ο ορισμός των ε, μη οικονομικών υπηρεσιών καθολικού συμφέροντος λοιπά, Είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ και χρόνια γιατί ο καθένας από εμά έχει μια διαφορετική κουλτούρα για τις δημόσιες υπηρεσίες. Όμως εμείς σήμερα βιώνουμε μια κρίση ταυτόχρονα που μας οδηγεί να αλλάξουμε στα κεφάλια μας όλοι μας αυτό το οποίο είχαμε ως ιδέα καταρχήν και αυτό μπορεί να μας επιτρέψει να ανοίξουμε τις ε, απόψεις μας. Εσωτερική αγορά λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιωτικό τομέα, τον δημόσιο τομέα, τους πολίτες και το δικαίωμα και, και το δίκαιο του ανταγωνισμού, μπορεί να μας οδηγήσει μεσοπρόθεσμα να βρούμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε αυτήν την εσωτερική αγορά για να αντιμετωπίσει. Τώρα κοιτάστε, εγώ σοσιαλίστρια είμαι, αλλά πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μου γίνεται συζήτηση για την αποπαγκοσμιοποίηση που εγώ την, βρίσκω ηλίθια. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να συζητήσουμε για την παγκοσμιοποίηση ως ένα τρόπο καλύτερης συμβίωσης. Ευχαριστώ λοιπόν Αντώνιο. Η εσωτερική αγορά βρίσκεται μέσα στις λεκάνες απασχόλησης που θα πρέπει να διατηρήσουμε και να δημιουργήσουμε και τις, το νέο εργατικό δυναμικό της αύριο. Ευχαριστώ κύριε σε κυρία Κοράτσα. Ευχαριστώ τον Αντώνιο, διότι είπε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, να προωθήσουμε την αποτελεσματικότητα της αγοράς και την καινοτομία. Συμφωνώ με τον Ανδρέας και τον Μάλκομ, διότι δεν πρέπει να ξαναρχίσουμε τη συζήτηση που είχαμε για την ενία εσωτερική αγορά. Η επικουρικότητα είναι ο σωστός δρόμος, άρα ας μην μπούμε από την πίσω πόρτα με αυτούς τους νέους ορισμούς προσπαθώντας να ορίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό με βάση τα όσα προελέχθησαν για την εσωτερική αγορά. Ο Ανδρέας το άρθρο 14, για το άρθρο 14 είπε ότι η νομοθετική πρόταση δεν είναι η σωστή. Μιλάμε για αποτυχία λειτουργία της αγοράς στην παράγραφο 1. Και στην παράγραφο 4 δεν έχει νόημα να μιλάμε για σαφείς διαφορές μεταξύ ε, υπηρεσιών οικονομικού και μη οικονομικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάιλερ τέλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που παίρνω το λόγο μετά από την ε, συνάδελφο, διότι εδώ πιστεύω ότι βασιλεύει μία μεγάλη διαμάχη και όλα αυτά τα ωραία λόγια που χρησιμοποιούμε δεν θα μας βοηθήσουν να τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Όταν υπάρχει μια αγορά ε, η οποία αποτελεί τη βάση για τόσο πολύ μεγάλη φιλελευθεροποίηση, εμείς είμαστε υπέρ της ρύθμισης και για τα οικονομικά έτσι συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει και μια ευρωπαϊκή συνένεση ότι και ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία στο παρελθόν έγινε υπερβολικές ε, απελευθερώσεις στις ε, αγορές. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα ε, αρχής. Και σωστά το είπε και ο Αντώνιο, αλλά το τόνισε και η Μπερναντέτ. Θεωρούμε ότι και η αγορά οφείλει να υπακούει σε κανόνες. Θυμούμε, και το προσθέτω στο τελευταίο σχόλιο, όταν συνέταξα την έκθεσή μου για τις κοινοπραξίες ιδιωτικού και δημοσίου τομέας, όπου όλοι θεωρούσαμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου πραγματικά τα πάνε καλά και υπάρχουν άλλες που πηγαίνουν άσχημα. Και είναι και κακά σχεδιασμένες και προκάλεσαν ζημιές. Όμως, ανεξαρτήτως αυτού, επιτρέπουμε να λαμβάνονται οι αποφάσεις επιτόπου και επιμένουμε μόνο στην τήρηση ορισμένων ελαχίστων ποιοτικών απαιτήσεων και θυμάμαι ότι ναι, οι συντηρητικοί χριστιανοδημοκράτες εννοώ τώρα θεωρούσαν, δεν δέχτηκαν την πρότασή μου όπου είχα πει δηλαδή ότι μια επανακοινοτικοποίηση μπορεί στην ουσία να είναι και πολύ σκόπιμη. Βεβαίως δεν περιλήφθηκε τελικά στην, στην έκθεσή μου. Τι έγινε τα τελευταία πέντε χρόνια και εδώ δυστυχώς οφείλω να σας αντίπω στην Γερμανία Υπάρχουν πολλές επανακοινωτικοποιήσεις επιμέρους έργων όπου αντίθετα με τη Μεγάλη Βρετανία έγινε πράγματι μια επανακοινωτικοποίηση και διεξάγεται συζήτηση τώρα και σε ομόσπονδα κρατήδια με κυβερνήσεις χριστιανοδημοκρατικές που σκέπτονται και πολύ σοβαρά εάν ίσω οι διάφορε διοικητικές περιφέρειες, μικρέ, μεγάλες κλπ, να επαναγοράσουν τμήματα ε, ε, επιχειρήσεων κοινή ωφελία τα οποία είχαν πωλήσει ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν νέες υπηρεσίες στους πολίτες. Επομένως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, όχι νέα ιδιωτικοποίηση, Και βεβαίως, όπως είπα, επανάκτηση των ε, τμήματων αυτών από τις κοινότητες, από, την, ε, από τις ε, διάφορες περιφέρειες. Εγώ είμαι πέρα αυτής της εξελίξεως, διότι οι μεγάλες απελευθερώσεις των αγορών οδήγησαν τελικά σε ζημία όλων και για την συλλογή των απορριμμάτων για παράδειγμα και για την υδροδότηση και για θέματα υγείας. Σε πολλά από αυτά σημειώθηκαν πολύ σημαντικές ελλείψεις μετά από αυτή την κίνηση. Θα παρακαλέσω τώρα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εκπροσώπο της με το δυσπρόφερτο όνομα, να λάβει το λόγο για να σχολιάσει τα όσα άκουσε και μετά θα δώσω τον λόγο στον καθηγητή Κιωτικάμπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήταν χρήσιμο ίσως να θυμίσουμε το πλαίσιο και το στόχο της μεταρρύθμισης των κανόνων για τις γενικές οικονομίες. υπηρεσίες ε, για τις υπηρεσίες ε, γενικού οικονομικού συμφέροντος εδώ δεν πρόκειται ούτε για ιδιωτικοποίηση ούτε για τίποτα άλλο. Μιλάμε εμείς για το πότε μπορούν να χορηγούνται αποζημιώσεις ε, στις, για τις δημόσιες υπηρεσίες. Η νομική βάση της πρότασης της Κομισιόν είναι το άρθρο 106 και όχι άλλο άρθρο της συνθήκης. Οι στόχοι αυτής της μεταρρύθμισης εξαγγέλθηκαν τον Μάρτιο. Πρώτος στόχος είναι η, διευ... διευκρίνηση συνενετική θέση. Υπάρχει βέβαια ένα όριο της, της Κομισιόν, δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται σεβόμενοι την ομολογία του δικαστηρίου. Αλλά φυσικά η Κομισιόν θα κοιτάξει να ξεκαθαρίσει όσο το δυνατόν περισσότερο ποιοι κανόνες εφαρμόζονται, όπως επίσης ε, και να εξηγήσει τι εστί η οικονομική υπηρεσία, τι μη οικονομική υπηρεσία, τι υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος όλους τους όρους δηλαδή που χρειάζονται για να ερμηνευτούν αυτοί οι κανόνες. Θέλουμε να έχουμε πιο διαφοροποιημένους κανόνες που να μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε υπόψη την μεγάλη ποικιλότητα των υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος αλλά και τις επιπτώσεις τους στον ανταγωνισμό ενδοκινοτικό ανταγωνισμό για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος θέλουμε να απλουστεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους κανόνες αλλά για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος με πολύ μεγάλες επιπτώσεις και που έχουν στην ευρωπαϊκή οικονομία θα πρέπει να δούμε τι αντισταθμίσεις θα έχουμε τόσο στον ανταγωνισμό αλλά και στη δημιουργία κινήτρων ούτως ώστε αυτές οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος να χορηγούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Δεν θα κάνουμε ένα τεστ αποτελεσματικότητας. Αλλά όταν μία, υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος χορηγείται σωστά, δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση. Καλούμε λοιπόν τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Εμείς ασχολούμαστε με τη σύνταξη των κειμένων αυτών, θα τους δημοσιοποιήσουμε σύντομα και θα διαβιβάσουμε στα άλλα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτό μας βοήθησε ιδιαίτερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως αυτό θα αντικατοπτριστεί και στη γνωμοδότησή μας. Ο εισηγητής θέλει να μας πει κάτι τελικά και να μας υπενθυμίσει το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρες. Δεν ε, πίστευα να μιλήσουμε για το θέμα σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικών επιστημών δηλαδή, κάτι το οποίο έγινε και με μεγάλη ε, χαρά διαπίστωσα ότι εκφράστηκαν πολλές απόψεις. Νομίζω ότι οι παρατηρήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες Υπάρχουν σημεία στα οποία δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Δηλαδή η απόφαση Altmark είναι μία απόφαση που μας σημάδεψε όλους. Μιλάμε επίσης για υπηρεσίες οικονομικού και μη ενδιαφέροντος. Μιλάμε για θέματα ανταγωνισμού. Επίσης συμφωνούμε σε σχέση σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τη διαφοροποίηση ε, κεντρικού κυβερνητικού επίπεδου, περιφερειακού και τοπικού. Εκεί που υπάρχουν διαφορές στην επικουρικότητα δηλαδή, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το όλο ζήτημα συγκεντρωτισμού, δηλαδή κεντρικής διευθέτησης. Φυσικά τα κράτη-μέλη διευθετούν το θέμα καταρχήν, διότι υπάρχουν αναταράξεις και ειδονισμοί. Δηλαδή υπάρχουν νομοθεσίες που αποκλίνουν και θα πρέπει να οριοθετηθούν. Αυτό δεν σημαίνει, Μάλκομ, ότι προσπαθούμε να εισαγάγουμε νέους ορισμούς. Η Επιτροπή ήταν σαφής ως προς τη ε, νεοριθέτηση των ορισμών. Θα ήθελα να τονίσω τον ποιοτικό ορισμό της Επιτροπής με αυτό το διάγραμμα σε σχέση με τα κοινά στοιχεία που υπάρχουν μεταξύ υπηρεσιών οικονομικού ενδιαφέροντος ή μη οικονομικό. Πρόκειται για ένα σαφές, σαφέστατο διάγραμμα. Γι' αυτό ε, λυπάμαι, αλλά δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε αυτό το άλοθη της επικουρικότητας θα πρέπει να ασχοληθούμε με κοινά θέματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα ζητήσω από το Μάλκομ να σας αποκαλύψω το εξής εξής. Ε, έμαθα πάρα πολλά από το Μάλκομ. Συζητάμε αυτά τα θέματα διαχρονικά και δεν έχουμε φτάσει σε ένα συμπέρασμα. Τώρα θα πρέπει να εκινήσουμε με μία νέα περίοδο, με μια νέα, σε μία νέα δεκαετία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επίτροπη. Η Επιτροπή ήταν απόλυτα σαφής και όπως είπε και ο Πρόεδρος ε, έθεσε το υπόβαθρο της συζήτησης, δηλαδή μας έδωσε όλα τα συμφραζόμενα. Μιλάμε για το άρθρο της νομικής βάσης, δηλαδή το άρθρο 106. Και βέβαια Βεβαίω ε, δεχόμαστε και την πάγια νομολογία του 10. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά όλων. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. θα συνεχιστεί η συζήτηση. Είναι η πιο, από τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις που με απασχόλησαν τελευταία δεκαετία, που με συνάρπασαν. Στις 2 Σεπτεμβρίου έχουμε την υποβολή ε, τροπολογιών γιατί θα πρέπει να ψηφίσουμε στις 19. Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τη γνωμοδότησή μας στις 4 ε, Οκτωβρίου και γι' αυτό η, η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων έχει κάπως καθυστερήσει. Θα πρέπει όμως να συνεισφέρουμε εμείς τώρα. θα υποβάλω και εγώ τροπολογίες, όπως και πολλοί άλλοι, και θα ψηφίσουμε στις 19 μιλώντας ε, για τους συμβασμούς. 19, 19, 19 Σεπτεμβρίου, εντάξει, ευχαριστώ, λέει ο κύριος Ντεκάμπος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες και τους ε, διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Σας ακούμε πολύ καλά και όχι, ως και όχι όπως κατά την πρώτη ώρα των εργασιών. Αύριο θα αρχίσουμε στις 9, θα μιλήσουμε σχέσεις, θα συζητήσουμε για τις σχέσεις μας με την Κίνα. Μετά έχουμε μία σειρά ε, ψηφοφοριών, να έχετε την ηλεκτρονική σας κάρτα. Μετά έχουμε ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις για την περιαγωγή, ενδιαφέρουσες μελέτες που θα ε, παρουσιαστούν και το απόγευμα θα αρχίσουμε με μια νέα νομοθετική πρόταση για τα δικαιώματα πνευματικών δικαιωμάτων. Και εδώ υπάρχει μια μελέτη, θα σας δω αύριο. Χαίρετε.